Κυρίες και κύριοι, καθίστε σας παρακαλώ. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, δημόσια πλέον συνεδρίαση. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους και τους παρόντες. Ελπίζω να περάσετε καλά το καλοκαίρι, να ξεκουραστήκατε και τώρα συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Τα επόμενα 75 λεπτά θα είναι αφιερωμένα στις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον κύριο Χάβιστο. Αγαπητέ Πέκα, καλωσορίσατε στην Επιτροπή Εξωτερικών. Χιβεπέιβε, όπως το λέτε και στα φιλανδικά. Καλά, το κατακρεώργησα. Ε, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ για τους συναδέλφους που εκλέγονται για πρώτη φορά ήθιστε στην αρχή της Προεδρίας να έρχονται οι Υπουργοί και να παρουσιάζουν το πρόγραμμα της εκάστοτε Προεδρίας για το επόμενο εξάμεινο. Η Φιλανδία λοιπόν ανέλαβε τη σκητάλη της Προεδρίας στα μέσα του έτους, αλλαγή σκητάλης και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν είναι εξαίρεση η σημερινή συνεδρίαση. Εμείς ε, ορίζουμε εισηγητέ ε, αυτό τον καιρό για τα βασικά θέματα. Ε, θέλω να καλωσορίσω και την μόνιμη αντιπρόσωπο της Φιλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργέ, η Επιτροπή μας σίγουρα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί νομοθετικά και πολιτικά με την Προεδρία σας για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα υπόλοιπα βασικά πολιτικά ζητήματα και προκλήσεις. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή στο Ελσίνκι και σήμερα το μεσημέρι εδώ και είμαστε πεπισμένοι ότι η Φιλανδική Προεδρία θα ε, εκμεταλλευτεί και θα αξιοποιήσει την πραγματογνωμοσύνη της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πείρα που έχει ε, σε ζητήματα διαμεσολάβησης για την ε, πύληση διαφορών και τις ειρνευτικές προσπάθειες. Θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων στη συνέχεια ε, έξι παρατέταρτο θα πρέπει να φύγει ο Υπουργό γιατί έχει άλλε ανηλυμένε υποχρεώσει. Έχετε και πάλι το λόγο, αγαπητέ Πέκα, παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, David. Ε, ε, Σα ευχαριστώ που επισκεφτήκατε και τη Φιλανδία. ξέρω ότι θα έρθουν και άλλοι βραβευτέ. είστε όλοι καλοδεχούμενοι βεβαίω αυτή τη στιγμή είναι και καλό ο καιρό, λέει ο πρόεδρο. Έω τώρα, έω τώρα, λέει ο υπουργό, ε, δεν μπορώ να σα εγγυηθώ τίποτα. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια σε όλου. Έχει ξεκινήσει μια πολύ σημαντική δουλειά ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικότερα ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίω ε, και στα πλαίσια τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εμεί θέλουμε να έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία μαζί σα. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τι απόψει σα, τι συμβουλέ σα κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα ο ρόλος ε, των Υπουργών Εξωτερικών, ο ρόλος του Υπουργού Εξωτερικού μάλλον είναι καινούργιο και για μένα. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνω, αναλαμβάνω αυτό το ρόλο. Ε, είχαμε εκλογές στην Άνοιξη, υπάρχει μια κυβέρνηση συνασπισμού πέντε κομμάτων. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, το καλοκαίρι είχαμε πολλή δουλειά ε, σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών, το θέμα της Ουκρανίας, ε, το θέμα της Βενεζουέλας με τη συμφωνία με την συνάντηση στο Περού. Ε, εκπροσώπησα την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Χαρτούμ, ε, στις ειρνευτικές συζητήσεις ε, και στην τελετή στο Σουδάν. Ε, πριν από κάποια χρόνια ήμουν μάλιστα και εκπρόσωπο, ειδικό εκπρόσωπο στο Σουδάν και στο Σουδάν και στο ήξερα το ζήτημα. Θα έχουμε λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα, μια ενδιαφέρουσα πενταετία σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε τη Φιλανδική Προεδρία. Πρώτα απ' όλα, Ξέρετε ότι είναι το σλόγγαν της Προεδρίας μας, μια βιώσιμη Ευρώπη, ένα βιώσιμο μέλλον. Η βιωσιμότητα προφανώς είναι ένα θέμα κλειδί για μας. Μιλάμε για την κυκλική οικονομία, αλλά μιλάμε και για κοινωνική και οικολογική βιωσιμότητα. Και είναι προφανές ότι το θέμα του κλίματος είναι στην καρδιά των προσπαθειών μας. Όταν δημιουργήθηκε ε, η νέα κυβέρνηση στη Φιλανδία, το θέμα του κλίματος ήταν πάνω πάνω στην ατζέντα, στο πρόγραμμά μας και πολλές άλλες κυβερνήσεις πλέον ε, έχουν αντιληφθεί ότι το θέμα της κλιματικής αλλαγής ε, είναι σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πετύχει τους στόχους της ε, του 2050 κλιματική ουδετερότητα. Εμείς, για μας ο στόχος είναι το 2035 στη Φιλανδία και προφανώς τα αισθήματα που αφορούν στο κλίμα ε, δημιουργούν πολλές προσδοκίες από αυτή την κυβέρνηση ε, θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή στενή συνεργασία με τον ύπατο εκπρόσωπο. Ξέρετε ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι κάπως διαφορετικός ρόλος της Προεδρίας. Εμείς παίζουμε έναν υποστηρικτικό ρόλο του του εκπροσώπου. Έχουμε μια σημαντική ε, εντολή να υποστηρίξουμε τον ύπατο εκπρόσωπο και οικονομικά και με τον προπολογισμό δηλαδή που θα έχει σε πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια. Υπό το φως βεβαίως του γεγονότος ότι πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Εμείς δεν είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά εξετάζουμε και το θέμα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις νέες απειλές, ε, υβριδικές απειλές. Ε, υπάρχει ένα κέντρο αριστείας στη Φιλανδία για τα υβριδικά αυτά ζητήματα και θέλουμε και εμείς να συνεισφέρουμε τις γνώσεις μας ε, στο θέμα αυτό. Στην, ε, στο σημερινό κόσμο ε, ξέρετε ότι οι διεθνείς σχέσεις αυτή τη στιγμή είναι τεταμένες και σε εμπορικό επίπεδο. Ε, εμείς θέλουμε να υπάρχει μια διεθνής τάξη που να βασίζεται σε σαφείς κανόνες, σε μια πολυμερή προσέγγιση υπάρχουν καταστάσεις όπως αυτή του Ιράν, η συμφωνία με τις χώρες του Μερκοσούρ ε, και βλέπουμε ότι η εμπορική πολιτική συνδέεται άμεσα ε, με την εξωτερική πολιτική. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό όταν θέτουμε στόχους σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Ένα από τα ζητήματα που η Φιλανδία έχει συμπεριλάβει στο κυβερνητικό πρόγραμμα αλλά και στο πρόγραμμα της Προεδρίας, είναι οι κοινέ αξίες μας. Τα κοινά συμφέροντά μας, να προστατεύσουμε τους, πολι... τους συμπολίτε μας, ε, να διαφυλάξουμε την παγκόσμια τάξη που αναβασίζεται σε κανόνε, αλλά και αξίε όπω τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη ελευθερία έκφραση, όλε αυτέ οι κοινέ αξίε που θεωρούμε ότι αποτελούν τη βάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτέ οι αρχέ δεν είναι διαπραγματεύσιμε. Είχαμε μια συνάντηση πριν από μερικές μέρες ε, στο Ελσίνκι. Ολοκληρώθηκε μάλιστα με τους εκπροσώπους των ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ε, γυναίκες περισσότερες από αυτούς, από τη Διεθνή Αμνηστία μεταξύ άλλων, που μπορούσαν να συναντήσουν λοιπόν και τους υπουργούς στο Γκίμνικ, μας είπαν τις εμπειρίες τους, ε, τις ιστορίες τους, τι μπορεί να κάνει και μας, ε, μας ζήτησαν τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι γνωστό ότι είμαστε φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και σε εθνικό επίπεδο. Η συνεργασία λοιπόν ε, τη Προεδρία μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ζητήματα αυτά σίγουρα θα είναι πολύ αποτελεσματική. Έχω ήδη αναφερθεί ε, στα κλιματικά ζητήματα. Εμεί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δείξει το δρόμο και διεθνώς για τα κλιματικά ζητήματα ε, δεν είναι μόνο ε, οι α, απαιτήσει, οι προποθέσει της συμφωνίας των Παρισίων και οι στόχοι που έχουν τεθεί. ξέρετε ότι υπάρχουν πολλέ χώρες διεθνώς που είναι διστακτικέ ε, για τα θέματα τα κλιματικά και να κάνουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Πρέπει λοιπόν εμείς να ασκήσουμε ε, μια επιρροή προς τις χώρες αυτές Θα πρέπει εμείς να είμαστε στην πρώτη γραμμή και να ηγούμαστε της προσπάθειας αυτή. Στην Φιλανδία έχουμε διαπιστώσει ότι και ο ιδιωτικός τομέας ή ο επιχειρηματικό κόσμος ε, τίνει πλέον να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτά, αυτή. Ο ιδιωτικος τομεας δηλαδή μας πρόχνει πλέον να κάνουμε περισσότερα. Μας λέει ότι η ευρωπη πρέπει να στην πρώτη γραμμή και τη τεχνολογική καινοτομία για τα ζητήματα αυτά εάν θέλουμε να φτάσουμε προς μια βιώσιμη, να πάμε προς μια βιώσιμη οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και να εξετάζουμε την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην οποία αναφέρθηκα. Ε, πρόσφατα είχαμε τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο. Ε, το συζητήσαμε και αυτό στο Γκίμνιχ. Πολλέ ε, ευρωπαϊκέ κυβερνήσει συμμερίζονται την άποψη ότι αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει στον Αμαζόνιο. Και εκεί πρέπει εμεί να παίξουμε ένα πιο ενεργό ρόλο. Ε, έχει να κάνει με τα δικαιώματα και των ε, ηθαγενών εκεί ε, και όσων ζουν στην περιοχή αυτή. Χάρηκα που και η κυρία Μογκερίνη ανέλαβε μια ισχυρή πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον κύριο Γκουτιέρες, τον Γενικό Γραμματέα των Εθνών, όταν μιλάμε λοιπόν ε, για το περιβάλλον, πρέπει να αναφερθώ και στο θέμα της Ακτικής, την περιοχή της Ακτικής. Ε, εκεί η Φιλανδία έχει δραστηριοποιηθεί εδώ και καιρό, είναι προτεραιότητά μας ε, και στα πλαίσια της Προεδρίας μας. Υπάρχουν εκεί πολλά και διάφορα συμφέροντα. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, υπάρχουν τα ζητήματα ναυσιπλοείας, σε μια ε, εποχή που αλλάζει το κλίμα ανοίγουν και νέοι δρόμοι ναυσιπλοεία, ε, νέες γραμμές τηλεπικοινωνίας και βεβαίω υπάρχει και στρατιωτικό συμφέρον εκεί. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέψει λίγο την προσοχή της και στο θέμα της τακτική και να έχει μια πολιτική και εκεί έτσι ώστε να μην αποτελέσει η περιοχή της ποτέ ε, αντικείμενο αντιπαράθεσης ή σύραξης. Ένα άλλο ζήτημα τώρα που έχει να κάνει με το πρόγραμμά μας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, ε, για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το ζήτημα της Αφρικής. Δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπονομεύει το τι συμβαίνει στην Αφρική, να το υποτιμά. Ε, σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο εμπορικό, πρέπει στην Αφρική να είμαστε περισσότερο παρόντες και οικονομικά και οικολογικά και κοινωνικά εκεί υπάρχει περιθώριο ε, μεγαλύτερης ε, συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης. Είναι δύο ισχυρά θεσμικά όργανα ε, που πρέπει να έρθουν πιο κοντά. Πρέπει να οικοδομήσουμε ε, δεσμούς, γέφυρες και να εξετάζουν, να, να βλέπουμε την Αφρική ως εταίρο, όχι να τους κοιτάζουμε αφιψηλού έχουμε και εμείς να μάθουμε από την εμπειρία των Αφρικανών. Θα ήθελα να αναφερθώ για άλλη μια φορά στην συμφωνία την ειρηνευτική στο Σουδάν. Ε, είναι πολύ σημαντικό να πετύχει αυτή η προσπάθεια. Στο Χαρτούμ υπήρχαν άνθρωποι που διαδήλωναν για έξι μήνες. Υπήρξε μια συμφωνία τελικά με το στρατό ε, για μια μεταβατική περίοδος, ενώ μέχρι πρόσφατα ήμασταν στα στα πρόθυρα της σύραξης. Υπάρχει γενικά αυτή η διάθεση που υπήρχε με την Αραβική Άνοιξη και ίσως, ίσως αυτό να μας δώσει τη λύση, μια βιώσιμη λύση για την ειρήνευση της περιοχής και αυτό θα το υποστηρίξουμε και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε απολύτως. Το Σουδάν δηλαδή θα μπορέσει ενδεχομένω να αποτελέσει παράδειγμα ε, για το πώς ανοίγει ο δρόμος προς τη δημοκρατία και την ειρήνη. Θα ήθελα στο τέλος της παρουσίασής μου να αναφερθώ στο θέμα των οικονομικών μέσων. Η Φιλανδία έχει μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία θέλουμε να υποστηρίξουμε ένα κοινό εργαλείο για την συνεργασία που θα δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Παράτυπη μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη, ξερώμαστε ένα πιο ευέλικτο όργανο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στι περιπτώσει αυτέ. Και τέλο, ένα ακόμα ζήτημα, το θέμα τη διεύρυνση. Στο Ελσίνκι είχαμε την ομάδα των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ε, με τη συμμετοχή και του Κωσυφοπεδίου ε, εμείς στη Φιλανδία θεωρούμε ότι η διεύρυνση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορούμε ε, να διασπείρουμε αυτές τις αξίες, αυτά τα συμφέροντα, τα κοινά που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και δεν υπάρχει, δεν μένει ποτέ τίποτα κενό. Αν δεν κάνουμε εμείς κάτι στα Δυτικά Βαλκάνια θα κάνουν άλλοι. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουν οι πραγματεύσεις αυτές ε, διαπραγμάτευση με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Ε, είναι ένα σημαντικό βήμα για την Ένωση. Ε, επικεντρωνόμαστε στη συζήτησή μας, αυτή τη στιγμή συζήτησή μα για στο Brexit, Ενδεχομένω χάνουμε κάποια από τα μέλη της Ένωση να έχουμε κατά νου όμως ότι υπάρχουν και μια σειρά από χώρε, μια ομάδα χωρών που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είχα να πω εγώ. Βλέπω ήδη ότι σηκώνονται κάποια χέρια, οπότε αναμένω τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Έχουμε περίπου 55 λεπτά για ανταλλαγή απόψεων. Θα πρότεινα να έχουμε ένα πρώτο γύρο εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων, να απαντήσετε εσείς και στη συνέχεια. Σε δύο γύρους. Δεν θα μπορούσα να δώσω το λόγο σε όλους που όλοι θέλουν να μιλήσουν. Πριν δώσω το λόγο στο Μιχαήλ Γκάλα, υποθέτω από το ΕΛΚ, θα ήθελα να πω το εξή. Ε, δύο σύντομα σχόλια. Πέκα, αναφέρθηκε στην πολιτική της Αρκτικής και ότι είναι προτεραιότητα της Φιλανδικής Προεδρίας θα ήθελα να σας συστήσω την έκθεση που εγκρίναμε εδώ στην Επιτροπή μας το 2017 για την πολιτική στην Αρκτική. Πάρα πολύ εμπεριστατωμένη, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και από τις σημαντικότερες εκθέσεις που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο για την Αρκτική για το 2017 πραγματικά ε, εξακολουθεί να ισχύει δύο χρόνια αργότερα το δεύτερο. Επειδή συναντηθήκαμε στο ε, Ελσίνκι, ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών με το, το, το φόρμα του Κίμνιχ, Είδαμε τον Ντάτσιτς, τον Σέρβο, να μιλάει έντονα με τον ομόλογό του του Κωσυφοπεδίου ε, τουλάχιστον συζητούν και μετά τις εκλογές της 6 Οκτωβρίου ίσως θα μπορέσουμε να τους ξαναφέρουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και οτιδήποτε κάνει και η Φιλανδική Προεδρία θα είναι πολύτιμο. Αυτά είχα να πω εγώ, ο κύριος ε, Γκάλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, στα φιλανδικά, ε, κύριε Κάβιστο. Αυτά περίπου. Εδώ σταματούν τα φιλανδικά μου. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζω στα γερμανικά. Ε, θα ευχηθώ στην Φιλανδική Προεδρία καλή επιτυχία. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για την επισκόπηση αυτή που μας ε, δώσατε. Θα ήθελα να τονίσω μερικές ψηφίδες. Αναφερθήκατε πολύ ε, στην προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω λίγο την εντύπωση ότι πολλές μεμονωμένες κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, στην υπόθεση του Hong Kong είναι πάρα πολύ διστακτικές για λόγους καιροσκοπικούς και οικονομικούς. Αλλά οι αρχές ε, τις οποίες εμείς πρεσβεύουμε είναι ανδιαφυσβήτητες και σίγουρα υποστηρίζουμε αυτό που συμφωνήθηκε πριν από 50 χρόνια. Δηλαδή μια χώρα δύο συστήματα. Και θα είχα το εξής ερώτημα. Εσείς δεν θα μπορούσατε ως Προεδρία να διατρανώσετε περισσότερο τις αξίες και τις αρχές μας. Γιατί αν πείτε εσείς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να βγει και να διαφωνήσει κάποια μεμονωμένη κυβέρνηση. Και να πείτε και στους Κινέζους ότι σεβαστείτε αυτό τουλάχιστον για αυτή την πεντηκοντά ετία μία χώρα δύο συστήματα, δηλαδή ελεύθερε εκλογέ στο Χονγκ Κόνγκ. Θα ήθελα να υποστηρίξω πάρα πολύ αυτά που είπατε σε σχέση με τη συνεργασία με την Αφρική. Έχω ασχοληθεί μακρόν με αυτό το θέμα και έχουμε μια αφορμή να ενισχύσουμε την Αφρικανική Ένωση. Είναι ενδιαφέρουσε οι εξέλιξεις για μια ζώνη ελευθερών συναλλαγών αφρικανική. Ερώτηση. Τι γίνεται όμως με τις συμφωνίες που έχουμε τις ΕΠΑ, ε, ε, οικονομικής ε, συνεργασίας και εταιρική ε, σχέσης. Αυτές θα υποκατασταθούν ε, από μια άλλη προοπτική, δηλαδή ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε με την Αφρικανική Ένωση μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ως μακροπρόθεσμο στόχο και τι θα κάνουμε στην πορεία προς τα εκεί, γιατί πολλά πράγματα ακόμα δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ενισχύσουμε το εμπόριο με την Αφρική και να το συνεχίσουμε. Δεν είπατε τίποτα για τη Ρωσία, παρόλο που έχετε τόσο μακρά χερσαία σύνορα με τη Ρωσία. Να θεωρήσω και να υποθέσω ότι η Φιλανδική Προεδρία θα συνεχίσει τη θέση που έχουμε για τη Ρωσία με τις κυρώσεις. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε και παρασκηνιακά στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ουκρανών κρατουμένων. Είτε πρόκειται για πολιτικούς κρατουμένους, για κάποιους ναυτικούς που έχουν συλληφθεί και κρατούνται. Εσείς που έχετε και καλές διασυνδέσεις με τη Μόσχα. Θα μπορούσατε να διαμεσολαβήσετε. Ε, ε, σταματώ εδώ, έχω και άλλα θέματα, να ρωτήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ Κάλε. Σοσιαλιστέ και δημοκράτε ο Τονίνο Πίτσουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, κυρία Πρέσβη, καλωσορίσατε ορίσατε στον Εκλογέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σα ευχαριστώ για τι εισαγωγικέ σα παρατηρήσει. Η εξωτερική δράση της Φιλανδικής Προεδρία και των προτεραιοτήτων τη. Ε, μιλήσατε για το κλίμα και για την ασφάλεια. Ε, είναι ευρέως γνωστό ότι η Φιλανδία διεθνώς ε, είναι πάρα πολύ ενεργή στην πρόληψη σειράξεων και στη διαμεσολάβηση. Ε, τώρα προτίθεστε να το ενισχύσετε αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, οι προτεραιότητές σας στην εξωτερική πολιτική συνήθως είναι συζητήσεις για τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται η ειδική ε, πλειοψηφία στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών και ε, ένα πιο ευέλικτο σύστημα για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, μιλήσατε για την πολυμερή ε, διάσταση και συνεργασία και για το εμπόριο. Πώς προτίθεται η Φιλανδική Προεδρία να ενισχύσει την αντοχή αυτού του συστήματος πολυμερού συνεργασίας γενικότερα, όχι μόνο στο εμπόριο. Και τέλος, συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπατε στο τέλος της παρουσίασής σας ότι η Φιλανδία θα βοηθήσει ε, ε, για μια προοπτική αξιόπιστη ένταξη των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, που είναι πολύτιμη περιφέρεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανία και η Κροατία, που είναι οι δύο επόμενες χώρες προεδρίας του Τρίου, έχουν την ίδια προτεραιότητα και θέλουμε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Ε, σας εύχομαι καλή επιτυχία καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ τον Νίνο. Ο κύριο από το Renew Europe. Thank you, uh, Minister, Σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ήμουν πρέσβη στη Φιλανδία και πρέπει να σας πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα ε, τις επαφές με τους ε, Φινλανδούς εκπροσώπους. Συνεχίζω λιγάκι στο ερώτημα το οποίο τέθη από τον συνάδελφό μου τον κύριο Γκάλα σχετικά με τις επαφές με τη ρωσική πλευρά. Ο κύριος Πούτιν επισκέφτηκε πρόσφατα τη Φινλανδία. Έχετε κάτι καλό να μας πείτε. Προέκυψε κάτι καλό από αυτή τη συνάντηση. Μήπως υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα της ε, Ουκρανίας, παραδείγματος χάρη ανταλλαγή φυλακισμένων ή ε, κάποια διευθέτηση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Προβλέπονται ε, κάποιες πρωτοβουλίες ενδεχομένω από δική σας πλευρά για να εξευρεθεί κάποια λύση. Και ένα άλλο θέμα εστιάζουμε στον Αμαζόνιο και έχουμε κάθε λόγο να το πράττουμε αυτό, αλλά και οι πυρκαγιές ε, στη Σερβία, αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλές, στη Σιβηρία με υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τελικά όμως δυστυχώς ε, δεν γίνεται τίποτα για αυτές τις ε, πυρκαγιές, δασικές πυρκαγιές. Ίσως να πιστεύετε ότι είναι πολύ πιο δαπανηρό να τις σβήσει κανείς από το να τις αφήσει απλά να μένονται και να συνεχίζουν δεν θεωρείτε ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή έτσι ώστε να προσφέρουμε κάποια ε, βοήθεια στην ε, Ρωσία έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές στη Συμβαρία ε, γιατί έχουμε κάθε λόγο να το πράξουμε αυτό. Μιλάμε για ιδιαίτερα εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές. Εκ μέρους των Πρασίνων, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Υπουργό στην Επιτροπή μας. Σας εύχομαι τα καλύτερα κατά τη διάρκεια της ε, Φινλανδικής Προεδρίας. Δείξατε πάρα πολλά θέματα, πολύ ενδιαφέροντα για τη διπλωματία, για το κλίμα, έρευνα και τεχνολογία, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Προσβλέπουμε σε πάρα πολλά και ελπίζουμε τα καλύτερα. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά το κλίμα. Ξέρω ότι αυτή είναι μία από τις ε, προτεραιότητές σας και θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα περισσότερο, πώς δηλαδή ακριβώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το θέμα της ε, διπλωματίας για το κλίμα. Ε, τι προτίθεστε να κάνετε, να εφαρμόσετε, μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος αυτού. Και υπάρχει άλλο ένα επίγον θέμα που πρέπει να δείξουμε είναι το Ιράν. Και θέλω να σας ε, συζητήσω ε, στις πρόσφατες ε, συζητήσεις που έγιναν να σταλεί μία αποστολή των ΗΕ στα στενά του Χορμούζ. Υπήρξαν κάποιες εξελίξεις. Ξέρω βέβαια ποια είναι η προσωπική σας άποψη σχετικά με αυτή την αποστολή. Δεν ξέρω τώρα ε, μήπως ε, μπορείτε να μας πείτε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Και θέλω να μας πείτε και μερικά περισσότερα πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς ε, καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας ήσασταν υπέρμαχος ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, υπάρχει ένα μοντέλο αυτό του Καναδά, θα μπορούσε ίσως αυτό να υιοθετηθεί ευρύτερα. θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσον προτίθεστε να δείξετε και αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν καλή τύχη στην Προεδρία σας. Ξέρουμε ότι ε, έχουμε καταλάβει ότι η αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγή είναι προτεραιότητά και εμεί σα υποστηρίζουμε. Μια προτεραιότητα όμω δεν, μπορεί, δεν πρέπει να μα ε, κάνει να ξεχνούμε άλλα προβλήματα. Θα αναφερθώ σε τέσσερα από αυτά. Το πρώτο είναι το θέμα των παράνομων μεταναστών. Η Φιλανδική Προεδρία δεν κρύβει τη βούλησή τη να προωθήσει σε κάτι που μοιάζει με μια αλλαγή αρμοδιοτήτων σε πέδο ασύλου. Και αυτό θα, είναι, θα έχει δραματικέ επιπτώσει. Λέτε λοιπόν ρητά ότι πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό τίτλο ό,τι αφορά το δικαίωμα ασύλου. Μπορείτε να μα το επιβεβαιώσετε αυτό. Ε, δεύτερον, σε επίπεδο πολιτική άμυνα, η φιλανδική κυβέρνηση θέλει να, να αυξήσει τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα τη στρατιωτική και την αντιμετώπιση των υβριδικών και ε, απειλών ε, στο διαδίκτυο ε, και, δεν, και αυτό γίνεται σε βάρος της αυτόνομης άμυνας της κάθε μίας χώρας ξεχωριστά. Μπορεί οι ευρωπαϊκές χώρες τελικά ε, να μπουν σε θανάσιμες παγίδες που θα μας θυμίσουν τον ψυχρό πόλεμο. Η Φιλανδική Προεδρία επίσης θέλει να προχωρήσει η ένταξη των χωρών Δυτικής, ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Αναφερθήκατε στη Βόρεια Μακεδονία ε, και ε, στην Αλβανία. Όμως υπάρχει και η Τουρκία. Η Τουρκία είπατε ότι είναι σημαντικό τέλο τη Ένωση. Θα συνεχίσετε ή θα σταματήσετε τι διαπραγματεύσει με την Τουρκία. Και τελευταίο ερώτημα. Η Φιλανδική Προεδρία αναφέρει ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ενιαία πολιτική απέναντι στη Ρωσία και στον τομέα των κυρώσεων. Αυτή η θέση που ουσιαστικά απαγορεύει οποιαδήποτε αλλαγή θέση απέναντι στη Ρωσία, μα ανησυχεί. Οπότε θα υποστηρίξω τον πρόεδρο Μακρόν κι εγώ για μια φορά, που ζητάει να αλλάξει θέση απέναντι στη Ρωσία. Εσεί πώ το βλέπετε αυτό. E Ευχαριστώ από την ομάδα ECR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Χάβιστο για την εισαγωγή του και του εύχομαι και εγώ κάθε επιτυχία στην Προεδρία, λέει ο κύριος Ρόισεν. Στο πρόγραμμά σας διαβάζω ότι δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στη διατλαντική συνεργασία και πολύ σωστά κάνετε. Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο αυτό ε, ε, η συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ για την ασφάλειά μας. Στο πρόγραμμά σας επίσης διάβασα ότι θέλετε περισσότερη ενότητα στην εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερα θέλετε να λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών με ειδική πλειοψηφία. Εκεί όμως διαφέρουν οι απόψεις μας. Πώς είναι δυνατόν να φτάνει σε ενότητα και ομοφωνία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι αναγκαστική ενότητα, επιβολή ε, της γνώμης των μεγάλων κρατών μελών. Δεν θέλουμε εμείς να πάρουμε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε είναι σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία ε, σε θέματα εξωτερικών και ότι θα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Άλλη ερώτηση. Μπορείτε λίγο να μπείτε σε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερα, ποιες είναι οι προθέσεις σας σε σχέση με το Ισραήλ ως Προεδρία συμφωνείτε μαζί μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι απολύτως στο πλευρό μιας χώρας ε, όπως είναι το Ισραήλ που απειλείται από τη Χαμάς, από τη Χισμολά, από το Ιράν το ίδιο. Παρακαλώ να μας πείτε τις προθέσεις σας. Και ένα τελευταίο. Σωστά αναφερθήκατε στα ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και ένα σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι η ανεξιθρησκεία. Είναι 73 χώρες παγκοσμίως όπου οι χριστιανοί διώκονται σοβαρά. Γνωρίζω ότι ε, το έχετε υπόψη σας, σας ερωτώ, ως Προεδρία θα το προωθήσετε για όσους ε, διώκονται για λόγους ε, θρησκευτικής πίστης και θα του δώσετε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην Προεδρία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράισεν. Και τώρα από την ΚΟΕ NGL, κυρία Βίλα Νουέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας και θέλω να σας ευχηθώ. Καλή επιτυχία. Ωραία ακούγονται τα λόγια σας για την ε, κλιματική επιτακτική πήγουσα κατάσταση, για την Αρκτική. Βεβαίως συμφωνούμε να υπάρξει ένα σαφές ε, στρατηγικό σχέδιο για την Αφρική, αν και θα χωρούσε πολλή συζήτηση το πώς θα γίνει αυτό. Θέλουμε να ρωτήσουμε το εξή: Μιλήσατε για τις διατλαντικές συμφωνίες, το διατλαντικό σύμφωνο. Σήμερα υπάρχουν οι πολιτικές ε, εκείνες συνθήκες για να συνάψουμε μια συμφωνία. Ο Τραμπ Δημοσίω είναι υπέρ τη διάλυσης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπονομεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Τι νόημα έχει να μιλήσουμε για μια συμφωνία με τι Ηνωμένε Πολιτείε και μια εξωτερική πολιτική πέρα από τα όσα κάνουμε. Είναι τώρα η στιγμή ε, απέναντι σε τέτοια ιδεολογία. Ε, τον Αύγουστο είδαμε να κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος Μακρόν σε 27 πρέσβεις λέγοντας ότι ε, ήταν ε, στρατηγικό σφάλμα να απομακρύνουμε τη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε κοντά μας τη Ρωσία. Εσείς τι γνώμη έχετε γι' αυτό και τι πιστεύετε για ε, τις μυστικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που μάθαμε τέλη Αυγούστου ότι ε, δημιουργήθηκαν στην Πολωνία. Ο νέος ύπατος εκπρόσωπος χρειάζεται ε, χάραξη νέας ε, πολιτικής για μεγαλύτερη αυτονομία και μεγαλύτερη στρατηγική ανεξαρτησία από τη Ρωσία, την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ. Και για να κλείσουμε τον πρώτο ε, γύρο, πάλι ο συνάδελφος από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον ε, κύριο Υπουργό για την παρουσία, λέει ο κύριος σας εύχομαι καλή επιτυχία. Δύο θέματα θα ήθελα να θίξω. Το πρώτο αφορά την αφορά στο πρόγραμμα της Προεδρίας της κοινές αξίες και το κράτος δικαίου. Όταν γίνεται λόγος για αξίες, εγώ που είμαι και συντηρητικός ευρωβουλευτής, ενοχλούμε πάρα πολύ γιατί δεν δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αξίες και αρχές. Και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι όταν συζητούμε για κράτος δικαίου και αρχές, δεν λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις αρχές που εμείς ορίζουμε ως κοινέ μας αρχές και αξίες. Μπορεί να γνωρίζετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το κράτος δικαίου αυτή τη στιγμή στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη. Και πώς μπορούμε εμείς να περιμένουμε όταν συζητούμε για διεύρυνση, να έρθουν νέες χώρες και να υπογράψουν αυτές τις βασικές μας αξίες ε, όταν δεν τις σέβονται τα νυν μέλη. Τι προτίθεστε να κάνετε ως Φιλανδική Προεδρία έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να σέβονται τις κοινέ αξίες αυτής εδώ της κοινότητας. Ε, πώς θα απατάξετε τη διαφθορά και πώς θα βεβαιωθείτε ότι όταν επιβάλλεται κυρώσεις αυτές δεν θα στρέφονται κατά των πολιτών των κρατών μελών αλλά κατά των κυβερνήσεων που φέρουν την ευθύνη. Το δεύτερο μου θέμα τώρα έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα και την ε, κοινωνική ένταξη που είναι και αυτά προτεραιότητές σας. Τα τελευταία χρόνια έχω διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από πολιτικό και οικονομικό διχασμό και δεν απολαμβάνουν εξίσου τα πλεονεκτήματα από την ενιαία αγορά όλοι οι πολίτες. Έχουμε τεράστιο μισολογικό χάσμα, ανεργία των νέων, ε, διαρροή εγκεφάλων από την περιφέρεια στο κέντρο, μαζική μετανάστευση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμείς θα θέλαμε να τη βλέπουμε ως ενιαία κοινή αγορά. Τι θα κάνετε εσείς, χρειάζεται μια νέα πολιτική συνοχής, χρειάζεται ένας επίτροπος ε, συνοχής, ε, χρειάζεται να μελετήσετε περισσότερο την ένταξη, την ενσωμάτωση. Πώς θα το χειριστείτε αυτό για να υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση στην κοινότητά μας. Ποια είναι τα μέσα και τα εργαλεία που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε και με ποιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρώτος ε, γύρος των ερωτήσεων. Ε, μπορείτε να απαντήσετε. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε κι άλλο ένα γύρο, γιατί εκεί θα ακολουθήσουν και πολλοί από τη Φινλανδία και από τη δική σα την πολιτική οικογένεια. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, ζητώ εκ των ε, προτέρων συγγνώμη, αν δεν μπορέσω να μπω σε βάθος ε, στι απαντήσει που θα δώσω. Κύριε Γκάλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τέλεια φινλανδικά σα. Δείξατε το θέμα του Χονγκ Κονγκ. Αύριο το θέμα αυτό θα συζητηθεί και θα έχουμε και τον εκπρόσωπο από το Πεκίνο και από το Χονγκ Κονγκ με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανησυχίες αφορούν στο ότι οι συμφωνίες που υπάρχουν στηρίζονται από όλου του άμεσα ενδιαφερόμενους. Αυτό το θέμα θα υπάρχει στην ημερήσια διάταξή μας ε, καθ' όλη τη διάρκεια του ε, φθινοπόρου, αλλά ε, περιορίζομαι καταρχήν σε αυτό που σας είπα ότι θα αισθηθεί το θέμα αύριο. Μετά, Όσον αφορά τη θέση της Φινλανδίας σε σχέση με τη Ρωσία και αν υπάρχει κάτι που ενδεχομένω έχει αλλάξει, ε, θέλω να σας πω ότι ήμουν στο Τορόντο ε, σε αυτή τη συνάντηση όπου ο νέος πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε την πρώτη του εμφάνιση και αν ακούσει κανείς πολύ προσεκτικά αυτά που λέει ο Ουκρανός πρόεδρος, εκείνος μίλησε για τον μη αποκλεισμό τη συμπερίληψη της Ανατολικής Ουκρανίας στην Ουκρανία. Μίλησε για ένα οικονομικό πακέτο προς τον Ντομπάς και την Ανατολική Ουκρανία. Μίλησε για το ανθρωπιστικό στοιχείο και μετά είδαμε όχι μόνο γενικές εκλογές στην Ουκρανία αλλά και αλλού και τώρα πλέον στηρίζεται πλήρως αυτή η γραμμή του. Νομίζω ότι είναι οι πρώτες προσπάθειες να υπάρξει πλέον διάλογος ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα και αυτό πρέπει να το καλωσορίσουμε. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να ακολουθήσει την, ε, το δρόμο της συμφωνίας ε, του Μίνσκ. Εκεί στη συμφωνία αυτή αναφέρεται λεπτομερώς το τι πρέπει να γίνει. Ανταλλαγή φυλακισμένων, απόσυρση στρατευμάτων, τα γνωρίζουμε. Και βεβαίως κατά την άποψή μας εμείς μετά θα πρέπει να προβούμε σε θετικές κινήσεις ε, και να υπάρξουν θετικές εξελίξεις τη σχέση με τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα όπως, τα, ε, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία του Μίνσκ κατά τα άλλα. Ε, νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βγούμε από αυτό το δίλημα, να στηρίξουμε τη συμφωνία του Μίνς και να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει διάλογος ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία για αυτά τα θέματα και για το θέμα της Κρυμαίας. Ε, κατόπιν ετέθη ένα θέμα του αν μπορεί η Φινλανδία να διαμεσολαβήσει στο να στηρίξει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Προφανώς και αυτό είναι προτεραιότητά μας και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει περισσότερο σε τέτοιου είδου θέματα. Μιλήσατε για την πολιτική του να υπάρχει ειδική πλειοψηφία. Εμείς στηρίζουμε την άποψη του να επικρατεί η ειδική πλειοψηφία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γιατί, διότι μέχρι τώρα υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τοποθετήθηκε, δεν είχαμε συμφωνία, είτε ήταν ανθρώπινα δικαιώματα, είτε και άλλα. Εμείς απλά παραμένουμε σιωπηλοί, δεν είπαμε τίποτα, γιατί δεν τα βρίσκαμε μεταξύ μας. Και οι ε, πρέσβεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας λένε ότι κοιτάξτε αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα λύσετε στο κέντρο και όχι σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, γι' αυτό το λόγο εμείς ως Φιλανδία στηρίζουμε το, την αρχή της ειδική πλειοψηφία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, είτε είναι για ανθρωπιστικά θέματα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Για το οικονομικό πλαίσιο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ε, ε, σας είπα ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό χαρτοφυλάκιο για τέτοιου είδους θέματα οικονομικής πολιτικής. Κατόπιν, όσον αφορά την ε, προοπτική διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων, ετέθη το θέμα αυτό και εγώ νομίζω ότι υπάρχει θετική προσέγγιση αυτή τουλάχιστον της Επιτροπής του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων. Όμως ε, το θέμα που ετέθη εδώ είναι πώς μπορούμε να είμαστε σοβαροί στο να στέλνουμε ένα σωστό μήνυμα στις ετούμενες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το κράτος δικαίου, αν αυτά δεν τα εφαρμόζουμε εμείς οι ίδιοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, σοβαροί όσον αφορά τις ε, κοινέ αξίες μας μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να λέει κανείς σε κάποιον άλλον, να ακολουθεί κάποιους κανόνες, αν ο ίδιος που το λέει τους παραβιάζει. Το επόμενο ερώτημα που ετέθη αφορά στις δασικές πυρκαγιές ε, στη Ρωσία. Δεν έχουμε μόνο ε, φωτιές στην Αμαζόνιο, στη Βολιβία, έχουμε και στη Ρωσία. Η Φινλανδία, τουλάχιστον στις ε, διμερείς σχέσεις, έχει θείξει το θέμα αυτό επανειλημμένα εναντί των Ρώσων. Ε, δεν είναι το μόνο περιβαλλοντικό θέμα που έχουμε τη Φιλανδία. Έχουμε το θέμα των επικίνδυνων αποβλήτων. Επίσης, ε, το θέμα ε, του μαύρου άνθρακα στην Αρκτική, όπου αυτός ο μαύρος άνθρακας καλύπτει τους πάγους και αυτοί λιώνουν πολύ πιο γρήγορα. Υπάρχει και το θέμα των εκπομπών θείου και εκπομπών άνθρακα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά εάν εσείς ρωτήσατε το αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σχετικά με την ε, διπλωματία του κλίματος. Συναντήθηκα με τον κύριο Γκουτέρες ε, πριν από λίγες ημέρες ε, και ε, τώρα περιμένουμε πάρα πολλά από τη συνάντηση κορυφή για το κλίμα του Σεπτεμβρίου. Θα ενθαρρύνουμε και στηρίξουμε όλου να προβούν σε πραγματικέ δεσμεύσει ε, ε, σε αυτή τη συνάντηση κορυφή. Εμεί θα συμμετάσχουμε στο ανώτατο επίπεδο και ελπίζουμε το ίδιο να ισχύσει και για άλλε χώρες. Και παράλληλα στηρίζουμε του στόχους του 2050 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι κάποιε χώρε διστάζουν ακόμα. Εμεί προσπαθούμε να πείσουμε ε, το δικό μας τον πρόεδρο και τους αρμόδιους να στηρίξουν αυτά τα θέματα. Ε, εγώ συναντήθηκα ας πούμε και με τον Πολωνό Κάτοβιτσε. Ε, πραγματικά εντυπωσιάζομαι από το ότι η Βαρσοβία κάνει κάποια βήματα για να ξεφύγει από τον άνθρακα, αλλά υπάρχουν άλλες περιοχές όπου βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στον άνθρακα και εκεί πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα. Ε, κάνατε μία ερώτηση για το Ιράν, για τις συναντήσεις τύπου Γκίμνιχ ε, στην ε, Φινλανδία. Είχαμε τη δυνατότητα να συνεντώ με τον Υπουργό εξωτερικό Ζαρίφ που επισκέφτηκε τη Φινλανδία και τις ε, σκανδιναβικές χώρες πριν πάει στην Ε, Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί καταρχήν το Ιράν είναι κατά του να υπάρχει στρατιωτική επίδυση στα στενά του Χορμούς. Από την άλλη όμως λέει ότι αν δεν υπάρχει και απειλή ε, για την ασφάλεια τότε δεν υπάρχει και ε, το, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει στρατιωτική επιχείρηση. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις εκεί στην περιοχή Υπάρχουν και άγνωστες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Κανείς δεν ξέρει ποιος επιτίθεται. Ε, αν μπορούμε όλοι να αγγιηθούμε ότι ε, δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδου επιθέσεις στο μέλλον, πράγματι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν τέτοιου είδου επιχειρήσεις για την αύξηση της ασφάλειας. Με πάση περιπτώσει, αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση, να στηρίξουμε το Ιράν, να παραμείνει στην GCP ε, και ε, να μην παίζει με την ιδέα του εμπλωτισμού ε, υλικών γενικότερα. Θεωρώ ότι οι Ιρανοί δεν πρέπει να κατηγορούν την Ευρώπη. Εμείς κάναμε τα μαθήματά μας εισαγωγικά. Ε, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να επιδείξει μια ιστορία επιτυχίας και πρέπει να παραμείνουμε σε αυτήν. Ο κύριος Μαριάννη έθιξε το θέμα ε, των προσφύγων, των ετούντων άσυλο στην Ευρώπη. Ε, δεν θέλω απαραίτητα να προσθέσω και ένα στοιχείο, να πω ότι όλα αυτά αφορούν ε, κυρίως τη Μεσόγειο, αλλά ξέρετε, όταν συμμετείχα σε ε, μία συνάντηση στο Περού, σοκαρίστηκα βλέποντας ότι οι πρόσφυγες της Βενεζουέλας είναι η δεύτερη ή τρίτη μεγαλύτερη ομάδα που έρχεται τώρα στην Ευρώπη. Και οι γειτονικέ χώρες, Κολομβία, έχει 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Μιλάμε συνέχεια για τους Σύρους πρόσφυγες, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται στην Λατινική Αμερική. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αλληλένδετα είναι τα προβλήματα και όλες αυτές οι παραβιάσεις ε, της δημοκρατίας, ε, κυρίως από πλευράς Βενεζουέλας. Για την Τουρκία. Δεν αναφέρθηκα στην Τουρκία, διότι βεβαίως είμαστε λιγάκι απογοητευμένοι με τις εξελίξεις, ε, τις τρέχουσες εξελίξεις στην Τουρκία και το πώς η Τουρκία προσεγγίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στη Φινλανδία πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο διάλογος. Εγώ συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, είχαμε μια καλή συζήτηση και υπάρχει κάποια μορφή συνεργασία. Είναι κρίμα όμως που η Τουρκία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Κατόπιν νομίζω ότι απάντησα ήδη για το θέμα της ειδική πλειοψηφία και θεωρώ... μισό λεπτό. Να περάσω τώρα στο τελευταίο σχόλιο που αφορά στο θέμα της, ε, του, της κατάργησης κοινωνικών αποκλεισμών. Ε, τελευταία ερώτηση από τον Ούγκρο συνάδελφο. Πράγματι πρόκειται για την ανεργία των νέων, ε, μαζική μετανάστευση μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου άνθρωποι προσπαθούν να βρουν ε, καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Ε, αν κάνουμε τα πράγματα σωστά, σε επίπεδο περιβάλλοντος και μερικές φορές είμαστε αναγκασμένοι να αυξήσουμε παραδείγματος χάρη τον φόρο των καυσίμων, πρέπει να υπάρχει ένα είδος αποζημίωσης των φτωχότερων, των πλέον ευάλωτων, έτσι ώστε και οι παραβολικές μας πολιτικές να είναι βιώσιμες. Ίσως να μην έχουμε βρει όλες τις απαντήσεις σε θέματα κατάργησης κοινωνικών αποκλεισμών, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι διαπιστώσαμε ότι πρέπει να παραμείνει ενωμένη ε, η ήπειρο μας και να προσφέρονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε όλους. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Είστε έτοιμος για το δεύτερο γύρο. Είναι τόσοι πολλοί συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δύο λεπτά έκαστο για να προκάνουμε. Ο κύριο Κουπίλη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σα ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε. Έχω δύο ερωτήσει που μοιάζουν με προηγούμενε. Θα προσπαθήσω όμω ε, έτσι να τις ε, τοποθετήσω υπό ένα κάπως διαφορετικό πρίσμα. Ε, Εξηγήσατε πολύ καλά γιατί είναι τόσο σημαντική η διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια. Εάν δεν ενεργοποιηθούμε εμεί, θα ενεργοποιηθούν άλλοι. Είναι σαφέστατο. Το γνωρίζουμε και εμεί από την εμπειρία μα πώ γίναμε μέλη τη Ένωση και με την υποστήριξη τη Φιλανδία. Αναφερθήκατε επίση στην κατάσταση στην Ουκρανία. Πολύ σύντομα συμμετείχατε και στη διάσκεψη του Τωρόντο. Τώρα έχουμε μια νέα κυβέρνηση πολύ δυναμική κυβέρνηση εκεί, από ό,τι φαίνεται, είναι πέρ μιας ε, προσχώρησης, μια προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα μου είναι σαφές και απλό. Τι μπορεί να κάνει η Φιλανδική Προεδρία, πώς μπορεί να στείλει ένα μήνυμα προς τη νέα αυτή κυβέρνηση, προς τον Ουκρανικό λαό, ότι είμαστε κοντά τους διότι φαίνεται μακριά η οποιαδήποτε βέβαια ένταξη της Ουκρανίας, αλλά πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφερθήκατε στη Ρωσία νωρίτερα. Παρακολουθούμε πολύ στενά τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Πούτιν. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μόσχα. Όπου Ρώσοι, Μοσχοβίτες, τους αρνούνται πολύ θεμελιώδη και απλά δικαιώματα, να είναι υποψήφοι βουλευτές. Και, και αυ... διαδηλώνουν. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ένωση ή η Προεδρία για να υποστηρίξει τους ανθρώπους αυτούς που ζητάνε να προσπιστούμε ένα θεμελιώδη δικαίωμά Θα δώσω τώρα το λόγο σε έναν πρώην συνάδελφό σα, τον ε, κύριο Βενίξα, πρώην Υπουργό. Ευχαριστώ. Ε, λέει ο κ. Μίξερ, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα τη πολυμερής προσέγγιση έγινε αναφορά προηγουμένω. Ε, υπάρχει μια κατάρρευση ίσω ε, τη τάξη αυτή ε, τη πολυμερούς. Αυτό φαίνεται κυρίω στον εμπορικό τομέα, αλλά και αλλού. Και σε ό,τι αφορά την πρόληψη αντιπαράθεση και σύραξη και στην επίλυση αντιπαράθεση. η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε συμφέρον να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της πολυμερούς ε, προσέγγισης. Όμως ε, θα πρέπει να έχουμε μία ενωμένη και ισχυρή ενιαία φωνή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο, σε διεθνή φόρα. Δεν συμβαίνει όμως πάντα αυτό. Δεν λένε όλοι τα ίδια στα Ηνωμένα Έθνη ε, τα κρατη της Ένωσης για σημαντικά ζητήματα. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τη μετανάστευση, ε, ο καθένας λέει τα δικά του, ακόμα και σε συστήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το να φτάσουμε σε κοινή ευρωπαϊκή ε, θέση ε, είχαμε... Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό. Μπλοκαρίστηκε επειδή μια χώρα της Ένωσης είχε πρόβλημα διμερέα, διμερές με μια τρίτη χώρα. Ε, ίσως να πρέπει να έχουμε ενισχυμένη πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία για να παίρνουμε αποφάσεις στα ζητήματα αυτά. Θα ήταν μια λύση τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Προεδρία σας έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε πιο ενωμένα, με πιο ενιαία φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σβέν για τους πράσινους. Τώρα κυρία Φέν Κραμών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να, συμφωνήσω, να αναφερθώ στο που ανέφερε ο κύριος Κουμπίλιους για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ε, Υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις στην Ουκρανία ως τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποιες νέες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αναλυφθούν όχι μόνο σε επίπεδο κοινωνία των πολιτών, αλλά και από άλλες ομάδες στην Ουκρανία ε, και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Φιλανδική Προεδρία για να υποστηρίξει τέτοιου είδους ε, μια νέα ατζέντα, αν θέλετε, μεταρρυθμιστική όπως αυτή που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση. Αναφερθήκατε στη συμφωνία του Μίνσκ Αναφερθήκατε και σε μια νέα μορφή διαλόγου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εάν δείτε όμως από κοντά τι συμβαίνει, δεν υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Έκανε μια έκκληση ο κύριος και στον κύριο Πούτιν, ξέρετε και τι του απάντησε ο κύριος Πούτιν. Δεν υπήρξε καμία απάντηση. Καμία απολύτως. Ο κ. Κουμπίλη αναφέρθηκε στην εσωτερική κατάσταση στη Ρωσία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση σε επίπεδο ρωσικής κυβέρνησης, ε, στο καθεστώς του Κρεμλίνου. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κάτι για το ποιες είναι οι δικές μας επιλογές για να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στον βρυδικό πόλεμο της Ρωσίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την παρέμβαση σε εκλογές ε, της Ρωσίας. Είστε από την Βαλτική, και τη Βαλτική θάλασσα, γνωρίζετε ότι εκεί λαμβάνουν χώρα ορισμένες φορές γυμνάσια εξαιρετικά ε, προκλητικά, ε, άλλες προκλήσεις της Ρωσίας. Λοιπόν, ε, δεν είναι μόνο ένα θέμα του επόμενου διαλόγου, του επόμενου βήματος του διαλόγου με τη Ρωσία και βεβαίως η κατάσταση στη Συρία μας ανησυχεί. Κλείνουμε τα μάτια μας στο θέμα της Συρίας, διότι έχουμε παγιδευτεί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει τουλάχιστον να ξεκινήσουμε μια νέα πρωτοβουλία για να υποστηρίξουμε τους Σύριους πολίτες ε, και την Συριακή αντιπολίτευση. Ίσως να έχετε κάποια ιδέα και γι' αυτό. Ευχαριστώ. Πολύ αγαπητοί συνάδελφε. Και πάλι από το ΕΛΚ τώρα η κυρία Σάντρα Καλνιέτε. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Ε, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Αναμένουμε ανυπομονησία την Προεδρία σας υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα στα οποία δεν αναφερθήκατε, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντική, σημαντικά για την Ευρώπη και για τη Φιλανδία και για όλες τις χώρες ε, της Βαλτικής και αναφέρομαι στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Δεν αναφερθήκατε σε αυτό. Η Ουκρανία αποτελεί μέρος της εταιρικής σχέσης. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Μολδαβία, η Γεωργία, που έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια μεταρρύθμισης. Μια προσπάθεια αλλαγής. Χάρηκα, διότι στο Γκίμνικ ε, αναφερθήκατε στις υβριδικές απειλές και υπήρξε μια κάποια συμφωνία μεταξύ των Υπουργών για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα ακόμα πράγματα επ' αυτού και ένα από τα πιο διχαστικά ζητήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες της Βαλτικής είναι το θέμα του Nord Stream 2. Τέλος, για τα Δυτικά Βαλκάνια χαίρομαι ιδιαίτερα διότι αναφερθήκατε στην αναγκαιότητα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με δύο εκ των χωρών αυτών. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη το 2003 όταν τους υποσχεθήκαμε ότι ανοίγει ο δρόμος για την Ευρώπη για αυτούς και είναι ακόμα στον προθάλαμο. Και να πω και δύο λόγια για τις αξίες, για την Κίνα και τη Ρωσία. Πρόκειται για δύο σημαντικές χώρες. Και στις δύο αυτές χώρες υπάρχει κοινωνική αναταραχή. Τι μήνυμα έχετε εσείς να στείλετε ως Προεδρία προς την Κίνα, για το Χονγκ Κόνγκ, προς τη Ρωσία, ε, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κοινωνικά δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σάντρα. σοσιαλιστές και δημοκράτες, κύριε Σουμουτσέβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, με ενδιαφέρον άκουσα το σύντομο σχόλιο σας για την Αρκτική. Αναφερθήκατε στην ασφάλεια, στις τηλεπικοινωνίες, αλλά υπάρχουν βέβαιως και άλλα σημαντικά ζητήματα. Μεταξύ αυτών είναι η φυσική πόροι. Πώς θα σας φαινόταν να θεωρήσουμε ότι είναι παγκόσμια κληρονομιά, όπως είναι και η φυσική πόρη στα βάθη των ωκεανών. Ξέρω ότι αυτό είναι αμφιλεγόμενο, αλλά είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να κάνουμε κάτι. Αλλιώς μια μικρή ομάδα χωρών θα μοιράσουν όλο αυτό το πλούτο μεταξύ τους που υπάρχει στην Ακτική. Ευχαριστώ. Ακόμα μερικούς αντέχετε. Ωραία. Σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλά την κυρία Χάιντι Χάουταλα, την επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Καλωσορίσατε, κύριε Πρόεδρε, στην Επιτροπή μας. Πραγματικά, ε, αναφερθήκατε στην εδρία ε, σε όσους ε, αγωνίζονται για υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, φάνηκε αυτό. Πολύ συχνά είναι αναγκασμένοι να φύγουν από τη χώρα τους. Δεν μιλάμε για πρόσφυγες και για ετούντες άσυλο, αλλά χρειάζεται να φυγαδεύονται. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, επανεκατάστασης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον σύντομης φιλοξενίας σε κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ανθρώπους αυτούς, αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, θέλω να δηλώσω τον ενθουσιασμό μου για τα όσα είπατε για την εμπορική πολιτική, ότι η εμπορική πολιτική είναι τμήμα της εξωτερικής πολιτικής. Μετά από το φετινό καλοκαίρι και τα όσα είδαμε στην Νότια Αμερική, αυτό το έχουν καταλάβει πάντες, αλλά όχι μόνο και παντού. Θα πρέπει πραγματικά να αλλάξουμε τακτική σοβαρά. Ε, συγκεκριμένα, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει έτσι ώστε το εμπόριο να ευθυγραμμιστεί με τις δεσμεύσεις μας και τις υποσχέσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Χάιντι Χάουταλα. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η κυρία Σάντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, Υπουργέ, για τα σχόλια σας και να ευχαριστήσω γι' αυτά. Και θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα χρειαστείτε μάλλον ακουστικά. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί άκουσα με προσοχή αυτά που μας είπατε για τις προτεραιότητες φιλανδικής ε, προεδρίας και σε μεγάλο βαθμό συμμερίζομαι ε, τις απόψεις σας. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω με πόση ευκολία χειρίζεστε και αναφέρεστε σε διάφορα θέματα, ιδιαίτερα όταν μιλήσατε για τη δυσκολία που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφανθεί για κάποια από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική. Και πώς καμιά φορά η Ευρώπη έχει χάσει το τρένο της εξωτερικής πολιτικής λόγω αυτής της αδυναμίας ε, ε, λήψης ταχαίων αποφάσεων. Επίσης, μιλήσατε για ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών για να μπορούμε να παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις σε τέτοια θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θα ήθελα εδώ να τονίσω τη σημασία που δώσατε ε, στα θέματα του περιβάλλοντος και ε, στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, μιλήσατε και για τον Αμαζόνιο όπως πολύ ωραία είπατε, δεν είναι πρόβλημα ε, δασικών πυρκαγιών εκεί. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα κράτους δικαίου και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένα θέμα σεβασμού των δικαιωμάτων των ηθαγενών ε, αυτοχθόνων λαών στη χρήση γης και πώς σε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα το δικαίωμα στη ζωή αυτών των αυτοχθόνων λαών, τους οποίους αυτή τη στιγμή δολοφονούν στον Αμαζόνιο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί αγωνιστές, ε, ε, πρασπιστές των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων που δολοφονούνται. Και αυτό το ε, καταματηρούν διάφορα στοιχεία και αριθμητικά για τη Βραζιλία. Πολύ σωστά λοιπόν είπατε Υπουργέ ότι το εμπόριο είναι εκ των Ρόνου κάνευ στην εξωτερική πολιτική και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς φαντάζεστε να εξελίσσονται οι ε, συζητήσεις στη Συμφωνία Μέρκοσουρ και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για την υπεράσπιση και πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ε, διώκονται και παραβιάζονται στη Βραζιλία και στον Αμαζόν. Λοιπόν, έχουμε ακόμα τέσσερις ομιλητές. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Η Φιλανδική Προεδρία και η σχέση μας με την Αφρική βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό. Ε, εμείς τα στηρίζουμε όλα αυτά, αλλά τελικά αυτό που διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα που ενδιαφέρουν ε, τα ιεραρχεί σε σχέση με την Αφρική και με άλλες χώρες ε, και αυτά όλα τα εντάσσει ως ένα κίνητρο στη συνεργασία. Εσείς ε, πώς ακριβώς αξιολογείτε την ισότητα ε, των, της συνεργασίας και κατόπιν υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το πράγματι μας ενδιαφέρουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, κυρίως σε σχέση με τους πρόσφυγες ε, που έχουν εγκλωβιστεί σε κάποιες ενδιάμεσες χώρες. Ε, και δεν ξέρω αν μπορούμε να τους προστατεύσουμε όλους αυτούς ε, σε σχέση με τη διαδικασία χορήγηση ασύλου. Ένας υπουργό, ο οποίος σε αυτούς τους έξι μήνες τι ακριβώ μπορεί να κάνει για να προάγει το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα και ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιες εξ εκτέσεις αξιολόγησης ε, σε άτυπες ή επίσημες ε, σχέσεις με τρίτες χώρες για θέματα μετανάστευσης. Να αξιολογούνται καλύτερα και όλες οι εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης. Η κυρία Αρένα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Πρώτον, κάτι που αναφέρατε εσείς και δεύτερον κάτι που δεν αναφέρατε σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Ε, είναι ένα ευρύτατο πεδίο, δεν είναι εύκολο να τα καλύπτουμε όλα. Σε ό,τι αφορά τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική, συμφωνώ απολύτω μαζί σα όταν λέτε ότι χρειάζεται μια ε, πολιτική επίση όρη. Ε, ωστόσο, αν κοιτάξουμε τον δείκτη της ανθρώπινης ανάπτυξης, 24 χώρες που είναι ουραγοί, δηλαδή λιγότερο ανεπτυγμένες ως προς την ανθρώπινη ανάπτυξη, είναι αφρικανικές, 24 από τις τελευταίες χώρες. Και στις 50 τελευταίες είναι όλες οι αφρικανικές. Δηλαδή, επίση, όρει είναι δύσκολο να συνομιλεί με τις χώρες αυτές όταν είναι τόσο ασύμετρες οι καταστάσει η Ευρώπη συχνά μιλάει για την πρόσβαση στους πόρους, στην Αφρική, στον πλούτο, για τη μετανάστευση και για το περιβάλλον. Η Φιλανδική Προεδρία, εκτός από αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά, είναι πρόθυμη να συζητήσει θέματα ευθύνη των εταιριών, των επιχειρήσεων όταν έχουν πρόσβαση στο φυσικό πλούτο. Πώς μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνε για τα ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς μπορούμε να τα βάλουμε δίπλα στην ασφάλεια, για τη μετανάστευση, πώς μπορούμε να συζητήσουμε για την κινητικότητα των όσων αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Αφρική. Στο θέμα που δεν αναφερθήκατε είναι το μεσανατολικό. Ισραήλ-Παλαιστίνη. Τι θέση έχει η Ευρώπη σε σχέση με αυτό. Σήμερα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η Ευρώπη ανέκαθεν ήταν υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Αυτή τη στιγμή ε, ε, η λύση αυτή ε, υφίσταται πιέσεις και από την Ισραηλινή κυβέρνηση και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πώς θα προωθήσετε αυτή τη λύση των δύο κρατών. Merci. Miss Κυρία Σατούρη, κύριος, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ ε, για την ε, παρέμβασή σας. Θέλω και εγώ να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ για τη Φιλανδική Προεδρία. Και όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι από την ομάδα των Πρασίνων, συμμεριζόμαστε τους στόχους σας για την κλιματική διπλωματία. Προσωπικά κύριε Υπουργέ, θα σας ρωτήσω για την κατάσταση στη Λιβύη. Όπως γνωρίζετε ε, είναι απάνθρωπες οι καταστάσεις που επικρατούν ε, στους καταβλισμούς εκεί, στα κέντρα σύλλου, με αυθαίρετες ε, κρατήσεις, και ε, εμείς ε, προτιμούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, δίνουμε υπεργολαβία αυτή τη διαχείριση στη Λιβύη και περιφρονούμε τις δεσμεύσεις μας. Η Φιλανδική Προεδρία έχει βάλει στην καρδιά της εξωτερικής δράσης τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεκατάστασης φιλόδοξο. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποια είναι η δική σας προσέγγιση και του Συμβουλίου σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στους καταβλισμούς στη Λιβύη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τελευταίος ο κύριος Κέστερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για όλα αυτά που μας είπατε. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω σε αυτά που μόλις τώρα μας είπε ο συνάδελφος. Η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική, αυτό είναι κάτι που το υπογραμμίσατε. Αν δούμε όμω λιγάκι την κατάσταση στη Λιβύη, δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να ισχυριζόμαστε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τη υποτιθέμενη λιβική κυβέρνηση ε, γίνονται σεβαστά. Έχουμε καταβλισμού όπου οι άνθρωποι ε, βασανίζονται, υφίστανται βασανιστήρια σε απίθανες καταστάσεις. Και η κυβέρνηση της Λιβύης τα εκμεταλλεύεται όλα αυτά ε, έτσι ώστε οι άνθρωποι που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο τους συγκρατούν, δεν τους αφήνουν να έρθουν στην Ευρώπη. Ε, εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει λιγάκι να τα ξανασκεφτούμε τα θέματα αυτά στη σχέση μας με τη Λιβύη. Ε, κατόπιν σχέσεις ε, της Δύσης με τη Ρωσία έχει επιδεινωθεί η σχέση αυτή λόγω της ε, μονομερής καταγγελίας από πλευράς ΗΠΑ της συνθήκης EFR. Εγώ λοιπόν ερωτώ μήπως υπάρχει εδώ κίνδυνος και πάλι των πυρηνικών επανεξοπλισμών η Ευρώπη μήπως πρέπει κάτι να κάνει έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την επανεμφάνιση όλων αυτών των πυράβλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Ε, δεν ξέρω πόσος χρόνος απομένει για να απαντηθούν όλες αυτές οι ερωτήσεις, αλλά παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ξεκινάω με τη Μέση Ανατολή. Γιατί ξέρετε κάτι και προηγουμένως το ξέχασα, κατά λάθο, μου ξέφυγε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της ύπαρξης του. Αυτό είναι ένα θέμα που έδειξα παραδείγματο χάρη στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Για μας αυτό είναι καθοριστική σημασία ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να αισθάνεται απειλή ως προς την ύπαρξή του. Παράλληλα βέβαια καταδικάζουμε την, ε, τους παράνομους οικισμούς, ε, την επέκταση των οικισμών σε αυτή την περιοχή, ε, να μην εμποδίζει τη λύση των δύο κρατών όπως έχουμε συμφωνήσει. Και αυτή θα πρέπει να είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμέναμε μέχρι τώρα την πρωτοβουλία των ΗΠΑ για την ειρηνευτική διαδικασία, τίποτα δεν έγινε και έρχεται κάποια στιγμή που δεν μπορούμε πια να περιμένουμε μόνο κάποιος τρίτος να κάνει κάτι. Όπως λοιπόν πολύ καλά γνωρίζουμε, όλα αυτά έχουν άμεση σχέση και με τα σχέδια του Ιράν, ε, τα σχέδια για πυρηνικό ε, σταθμό. Ελπίζω, λύνοντας το πρόβλημα του Ιράν, θα υπάρχει χώρος και για μια πιο ασφαλή Μέση Ανατολή. Και ένα άλλο θέμα που ξέχασα προηγουμένως να δείξω, ε, το θέμα των ε, θρησκευτικών αξιών. Είναι αυτονόητο ότι όταν μιλάμε για ε, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προφανώς μιλάμε και για θρησκευτικά δόγματα, ομολογίες, οτιδήποτε είναι αυτά. Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους, το δικαίωμά τους να εκφράζουν τις απόψει τους και να καλλιεργούν τα πιστεύω τους. Ο κύριος Κομπέλιους έθεσε ένα ερώτημα πιο συγκεκριμένα για την κατάσταση στην Ουκρανία και το τι μπορεί να κάνει η Φινλανδική Προεδρία. Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να στηρίξουμε τον νέο πρόεδρο στην Ουκρανία, το νέο κοινοβούλιο, εμείς είμαστε η μεγαλύτερη, η σημαντικότερη εμπορική εταίρεια της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή. Ε, είναι λοιπόν απόλυτα σαφές ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή είναι και η απάντησή μου σχετικά με την ε, ανατολική γειτονία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά με τις χώρες αυτές σε οικονομικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα, ως προς την αντίδραση ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, ε, προφανώς αντιδράσαμε γέρος ε, και δεν είναι καλό ε, να μην μπορούν να υπάρχουν υποψήφοι για τις τοπικές εκλογές και για την Δούμα και κατανοούμε από πού ε, προέρχονται οι αντιδράσεις. Το θέμα της πολυμέρειας. Ε, Τέτοι προηγουμένως το θέμα των διατλαντικών σχέσεων. Πώς δηλαδή μπορούμε τις ε, διατλαντικές σχέσεις να τις διαμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην αποφασίζει απαραίτητα η άλλη πλευρά. Αλλά ξέρετε πρέπει να έχουμε υπομονή. Έχουμε πάρα πολλά κοινά συμφέροντα με τις ΗΠΑ και γι' πρέπει να είμαστε πολύ υπομονετικοί. Ε, εγώ δεν θα το αφαιρούσα το θέμα αυτό από τη δική μας την ημερήσια διάταξη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες θα παραμείνουν ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για θέματα κλιματικής αλλαγής και άλλα. Παρόλα αυτά πρέπει να διατηρηθούν οι σχέσεις μας. Ετέθη ένα ερώτημα σχετικά με την Ουκρανία αλλά και για τη Συρία. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Βεβαίως, όπως συμβαίνει πάντα, ε, εδώ περιλαμβάνεται και η Τουρκία, η Ρωσία, οι δυτικές δυνάμεις, η κυβέρνηση στη Ρωσία. Ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε πλέον όλοι είναι η κατάσταση του στον καταβλισμό Ανχολ. Ε, Επιτέλου, αυτό ήταν μια επιτυχημένη έκβαση ε, το θέμα του ISIS ε, και τώρα βλέπουμε δυστυχώς ότι τα παιδιά και οι γυναίκες ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες στον καταβλισμό Ανχολ. Και βλέπουμε επίσης ότι δυστυχώς διαδίδεται και η ιδεολογία του ISIS. Εμείς ακούμε όμως από την άλλη ότι στο Αφγανιστάν επανεμφανίζεται το ISIS και σε κάποιες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις στην Ασία, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επέτει ένα ερώτημα σχετικά με την Ανατολική γειτονία. Νομίζω απαντήθηκε αυτό το ερώτημα. Να σας πω λιγάκι και το τι είπαν οι Υπουργοί Εξωτερικών. Μιλήσαμε για παράνομη ε, χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, παραπλάνηση, ε, fake news, όλα αυτά τα θέματα τα οποία δεν είναι πια ε, και τόσο μοντέρνα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ καλύτερα όλες αυτές τις μεθόδους που παρισφρέουν τώρα στις κοινωνίες μας. Αναφερθήκατε και στον εγώ North Stream που αναμφισβήτητα επηρεάζει την κατάσταση στην Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για μας, ε, για τη Φιλανδία, εντάξει δεν μας αφορά γιατί δεν παίρνουμε ε, αέριο από τον αγωγό αυτό, το κοιτάμε περισσότερο από περιβαλλοντική σκοπιά, αλλά και από το πρίσμα της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων μας στην Ανατολική Γειτονία κύριος Σίνασεβιτς έκανε ένα ερώτημα σχετικά με την Αρκτική, ε, κατά πόσο ενδεχομένω θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι ε, φυσικοί πόροι. Ε, αυτά που υπάρχουν στο βυθό της θάλασσας. Δεν πρέπει να υπάρχουν οι εκπομπές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα και δεν θα υπάρχουν αν μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα ορυκτά καύσιμα κυρία Χάουταλα έκανε ένα ερώτημα το τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά κάποιον τρόπο να, τους, να υπάρχει ένας μηχανισμός προστατευτικός. Νομίζω ότι είναι καλό να ε, σκεφτούμε το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Και σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες, κοιτάξτε, για το Μερκοσούρ οποτεδήποτε μιλάμε για τη Βραζιλία, για τις ε, πυρκαγιές, μερικοί λένε δεν θα πρέπει να δεχτούμε τη συμφωνία Μερκοσούρ, αλλά όσοι πεστορίζουν το Μερκοσούρ λένε ότι υπάρχει συμφωνία του Παρισίων, υπάρχουν άλλες συμφωνίες και υπάρχει μία αρχή ότι δεν θα πρέπει να εισάγονται ε, ποσότητες κρέατος από περιοχές που αποψηλώθηκαν πρόσφατα. Ε, το περιβαλλοντικό στοιχείο εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί περισσότερο στις ε, συμφωνίες μας. Και αυτά είχα να πω και προς την κυρία Σάντος, που εσείς ε, και το θέμα της σχέσης ε, ανάμεσα στους υπέρμους ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτούς ε, που ασχολούνται με το περιβάλλον. Εγώ πρόσφατα ήμουνα μάρτυρας μιας τέτοιας αντιπαράθεσης ε, και πραγματικά βλέπουμε ότι πολλοί που είναι γηγενείς ε, και αγωνίζονται για το κλίμα, πολλοί εξ αυτών δολοφονούνται. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Η κυρία Στρίκτ έκανε ένα ερώτημα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θέματα της μετανάστευσης. Ε, θέλω να πω και κάτι που βρίσκεται στη ρίζα του προβλήματος, γιατί γίνεται ε, μιλάμε συχνά γι' αυτό. Οι οργανώσεις της Φινλανδίας ίσως είναι από τις λίγες που εργάζονται ε, στο, στην Ερυθρέα. Πράγματι, ε, είναι ένα θέμα αυτό που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά βλέπουμε και στη χώρα επιτόπου ανθρώπους που να λένε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να σπουδάσει κανείς και υπάρχουν εκεί οργανώσεις που διδάσκουν τους δασκάλους. Μερικές φορές ε, αυτά ε, τα αίτια, ίσως να χρειάζονται και κάποια βοήθεια έτσι ώστε και να μπορούν οι πολίτες ε, να κάνουν τις σωστές επιλογές. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Έρχομαι τώρα στην τελευταία μου παρατήρηση. Η κυρία Ρένα μίλησε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Το θέμα είναι κρίσιμο, ε, πρέπει να μας απασχολήσει όλους περισσότερο. Για τη Μέση Ανατολή ήδη απάντησα, ο κύριος Σατούρη έθεσε το θέμα της Λιβύης, Πράγματι θα πρέπει να στηρίξουμε το ειρηνευτικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι μια χώρα η οποία διολυσταίνει σε αυτό το δράμα του εμφυλίου πολέμου, ε, εκεί ε, αναπτύσσονται όλες οι μορφές ε, ανθρώπινου δουλεμπόριου, εγκληματικότητας. Ο κύριος Κιώστερ και εκείνος έθιξε το θέμα αυτό. Και τέλος, ε, το τελευταίο ερώτημα αφορά Ρωσία, Ηνωμένε Πολιτείε και πυρηνικά θέματα. Με ανησυχούν πάρα πολύ τι συμβαίνουν με τη συμφωνία INF. Ε, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δεν ξέρω αν ήμασταν ε, σε αυτή τη φάση τα πράγματα αυτά είναι διαφορετικά. Τώρα όμως θέλουμε όλοι να ξεφορτωθούμε τα πυρηνικά όπλα και άλλα όπλα μαζικής ε, καταστροφής. Ε, πρέπει πράγματι να ε, λογικευτούμε σε όλα αυτά τα θέματα. Το ίδιο ισχύει βεβαίω και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ακούσατε τι ερωτήσει μα, απαντήσατε, κάνατε και τα σχόλιά σα, Καλή τύχη, έχετε πολλή δουλειά μπροστά σα. Okay, Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, φτάνουμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα, στην μέσα διάταξη, το σημείο παριθμών 5, στην εισφορά της ΑΦΕΤ στην ετήσια δημοσιονομική διαδικασία για τον προπορισμό του 2020. Να θυμίσω ότι είναι η ίδια διαδικασία που ακολουθούμε κάθε χρόνο δύο διαφορετικά στοιχεία, έτσι, διαδικαστικά, η, το ψήφισμα της ΑΦΕΤ και οι τροπολογίες του προπολογισμού μετά από προτάσεις ε, του, μετά το σχέδιο προπολογισμού του, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει όμως αποσύνδεση των δύο διαδικασιών πλέον. Θα ψηφίσουμε αύριο πρωί για τις τροποποιήσεις, για τις τροπολογίες, ενώ μόλις την 1η Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε επί της γνωμοδότησής μας. Αυτά είχα να πω. Ο Μίχαλ Γκάλερ τώρα, ο εισηγητής, θα σας παρουσιάσει το σχέδιο εισήγηση και την προσέγγιση του σε ό,τι αφορά το θέμα των τροποποίησεων. Ευχαριστώ, Ντέιβιντ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο προπολογισμό ε, δεν είναι έτσι ένα τόσο σεξι θέμα προς συζήτηση, γι' αυτό είμαστε και λιγότεροι, αλλά κάποιοι γνωρίζουν ότι και στον προπολογισμό μπορούμε να προβούμε σε κάποιες αλλαγές. Ε, βλέπω εδώ και αριστερά και δεξιά κόσμο έχει. Στο κέντρο δεν έχει κόσμο, απλώς το αναφέρω. Ναι, κάποιοι, βλέπω κάποιους που λείπουν, για να το πω έτσι. Λοιπόν, ε, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τους και όλους τους από τις διάφορες πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία τους και την υποβολή τροπολογιών, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και το περιορισμένο χρονικό διάστημα που είχαμε με το καλοκαίρι. Ο προπολογισμό ε, είναι η καρδιά και η ραχοκαλιά των εργασιών μα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο εφόσον έχουμε του απαραίτητου πόρου θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε ε, των πολιτών μα. Οι προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλέ. Και οι πολίτε δικαίω αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποτελεσματική, να είναι δραστήρια και στην άμεση γειτονιά μας, αλλά και ως παγκόσμιος δράστης, ως παγκόσμιος παράγοντας. Ε, μετά το σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν του Ιουνίου και τη θέση του, του Συμβουλίου τον Ιούλιο, ήρθε η ώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας να ακούσει η φωνή μας ε, έτσι ώστε να υπάρξει κατάλληλη και αποτελεσματική χρηματοδότηση των εργασιών μας. Βεβαίως ε, έχω κάποιους συναδέλφους ε, που έχουν υποβάλει τροπολογίες που αρέσκονται στις δαπάνες. Ε, προσπάθησα να ακολουθήσω εδώ ε, την εξή προσέγγιση. Όταν έχει να κάνει με το επίκεντρο των εργασιών μας, τον πυρήνα των εργασιών μας, έχω υποβάλει τροπολογίες για να αυξηθεί ο προπολογισμό. Και όταν λέω πυρήνα εννοούμε σε νότια γειτονιά, ε, πολιτική γειτονία ανατολικά, ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν όμως είναι εκτός του πυρήνα των δραστηριοτήτων μας και είχαμε μια περίπτωση με μια τροπολογία από μία μόνο πολιτική ομάδα και που δεν αποτυπώνονται και στις ε, επιτροπές που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, αντίστοιχες ε, προτάσεις ε, τότε και εγώ δεν τα προωθώ. 11 λοιπόν τροπολογίε συμβασμού έχουν συμφωνηθεί, που μπορούν να γίνουν αποδεκτέ από όλου, πιστεύω, αφορούν σημαντικού τομεί πολιτική τη Ένωση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιου από αυτού πιο λεπτομερώ. Ζητούμε 10% ή 4,6 εκατομμύρια αύξηση στον προπολογισμό για τις ε, ε, αποστολές παρατηρητών στις εκλογές, διότι συνεισφέρουν στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ε, των κοινωνιών στην εκλογική διαδικασία ε, ενισχύοντας έτσι και άλλους στόχους εξωτερικής πολιτικής όπως παραδείγματος χάρη είναι η οικοδόμηση της ειρήνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα υποστήριζε ε, τις σχετικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί συναδέλφοι μας έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου αποστολές. Ε, Επίσης στο συμβιβασμό ζητάμε αύξηση της χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά το μέσο ε, εταιρική σχέση με τρίτες χώρες πάντα σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις, και τις ελευθερίες. Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων και ε, ευθυγράμμιση με κοινωνικό κεκτημένο στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στον τομέα της μείωσης της φτώχειας, επίσης αύξηση της χρηματοδότησης ε, ε, για την ε, Παλαιστίνη ζητούμε αύξηση του κεφαλαίου που έχει να κάνει με την οικοδόμηση εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση ε, των αντιπαραθέσεων και σε ό,τι αφορά την εταιρική σχέση με την Ανατολή και σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση λόγω των εξελίξεων στην περιοχή μεταξύ των οποίων βεβαίως τη σύραξη στη Συρία, στη Λιβύη, την εμπόλεμη κατάσταση, ε, η σύραξη αυτή καθ' αυτή και οι μεταναστευτικές ροές, οι ροές των προσφύγων. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις προσπάθειες ε, σταθεροποίησης των χωρών αυτών. Ζητούμε λοιπόν αύξηση της τάξης του 10%, 63 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή υπάρχει μια επιδείνωση και στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης ό,τι αφορά ζητήματα ασφάλειας θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της οικοδόμησης εμπιστοσύνη με τους ανατολικούς εταίρους μας. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για να προωθήσουμε τη δημοκρατία ε, και την σταθερότητα στην περιοχή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά βεβαίω την Ουκρανία, αλλά και τα, την εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική ε, Ουκρανία. Εκεί ζητούμε 7% αύξηση, 9% εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Πιστεύουμε ότι είναι ισορροπημένες ε, οι προτάσεις μας. 900.000 ευρώ συγγνώμη αύξηση για την Ανατολική Ουκρανία. Ε, υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που έχουν να κάνουν με ζητήματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς μας. Κατά τη γνώμη μου όμως, η ΑΦΕΤ πρέπει να συζητήσει και να ψηφίσει αυτές τι τροπολογίες που έχουν να κάνουν με ζητήματα που σχετίζονται με ζητήματα δικά μας. Κάποια άλλε κάποιες άλλες ε, τροποποιήσεις, κάποιες άλλες όμως δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία πρόταση, πρόκειται για την τροπολογία 5296 που προτείνει στον Άλεφο Σάντος η Επιτροπή την εξέτασε ε, και έλαβε κακό βαθμό, C. Θα ήθελα να σας διαβάσω εδώ τι λένε οι υπηρεσίες της ε, Κομισιόν γι' αυτό. Λέγεται λοιπόν εδώ, η πρόταση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Έχει να κάνει με ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την πρόληψη, την, ε, την, πρόληψη και την καταπολέμηση της ε, ε ατιμορρησίας. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση διότι καλύπτεται ήδη από την εξής, ε, τις εξής ε, νομοθετικές δραστηριότητε. Το Ευρωπαϊκό ε, Εργαλείο για τα Δημοκρατία και τα Δικαιώματα, η Κομισιόν προτείνει το πεδίο αυτής της πρότασης να συμπεριληφθεί εκεί, στο Ευρωπαϊκό Μέσο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προσθέτοντας αυτές τις ε, δαπάνες στην αντίστοιχη δημοσιονομική γραμμή. Αυτό θα προωθήσει τις προσπάθειες πολέμηση της ατιμορρησίας για τα πιο σοβαρά εγκλήματα, ενισχύοντας και την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζοντας τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της κόσμιας στρατηγικής και της, ενισχυ... της ολοκληρωμένης προσέγγισης ε, στις κρίσεις και στις σειράξεις. Εντάσσεται αυτό και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την υποστήριξη ε, σε ό,τι αφορά τη μεταβατική ε, δικαιοσύνη, την, ε, το, το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο και δίνει μεγαλύτερη οτότητα στην προσέγγιση της Ένωσης ό,τι αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση της ατιμορρησίας ε, για, τα πιο, για τις πιο σοβαρές μορφές εγκλημάτων. Θα ήθελα να ζήσω από τον συνάδελφο, τον Σάντος, λοιπόν, κατά πόσο ε, μπορεί να αποδεχτεί να ακολουθήσουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κατά πόσο θέλετε παρόλα αυτά να ψηφιστεί η πρότασή σας αύριο, να τεθεί στη ψηφοφορία. Ε, εγώ θα μπορούσα να υποστηρίξω επί της αρχής αυτή την ε, τροπολογία. Βεβαίως ε, είναι πιθανό στη συνέχεια στους συναδέλφους της αρχης αυτη την τροπολογια Βεβαίω ειναι πιθανο στη συνεχεια στους τη της επιτροπης προπολογισμου να μην προχωρήσει Εάν όμως ακούσετε ε, την συμβουλή της Κομισιόν και ακολουθήσετε αυτή την οδό, ενδεχομένω να μπορέσει εκεί να βρεθεί μια λύση. Εν μια ακόμα τελευταία πρόταση, η τελευταία τροπολογία 5257, 5257 ε, έχει να κάνει Ε, στην αρχή είχαμε μια τροπολογία μάλλον μόνο με τα επιχειρήματα για τις εξελίξεις ε, σε ό,τι αφορά τις χώρες ε, διεύρυνσης κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στα εθνικά κοινοβούλια. Η μεταρρύθμιση αυτή, η περιτροποποίηση αυτή υπάρχει, όμως οι εμπειρογνώμονές μας, το δικό μας προσωπικό, αλλά και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης είπαν, ακούστε, είναι καλή αυτή η πρόταση, να εξετάσουμε το πώς εφαρμόζεται αυτά που αποφασίζουμε εμείς σε επίπεδο Εθνικών Κοινοβουλίων, θα μπορούσαμε με πολύ χαμηλό κόστος τις χώρες αυτές, ε, στις χώρες συνδεδεμένες με την Ένωση έτσι, και τις χώρες της διεύρυνσης, θα μπορούσαμε να προσλάβουμε τοπικά εκεί προσωπικό που να εξετάσει σε εθνικ, στα επίπεδα εθνικών κοινοβουλίων ε, με τις πολιτικές ομάδες, ε, τις κοινοβουλευτικές ομάδες ε, κατά πόσο τα συμφωνημένα εφαρμόζονται και προχωρούν. Και εκεί μπορεί να έχουμε μια αύξηση τάξη των 400.000 ευρώ. Αφορά 10 χώρες, έτσι. 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Τουρκία, την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Ιδιαίτερα βεβαίω στην Ουκρανία και στη Μολδαβία ε, έχουμε νέες κυβερνήσεις ε, που έτσι με ενθουσιασμό θέλουν να εφαρμόσουν αυτή την ατζέντα μεταρρυθμίσεων που έχουμε συμφωνήσει. Αύριο λοιπόν ε, στην ψηφοφορία θα υποβάλω μια προφορική τροπολογία για αυτή την αύξηση 300.000 ευρώ για να καλυφθεί αυτό το κόστος. Και καλό θα είναι οι συνάδελφοι να το υποστηρίξουν αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Μιχαήλ Γκάλα. Πριν δώσω το λόγο στους και οδησηγητές, θα ήθελα σύντομα να επανέλθω σε ένα σημείο που ανέφερε ο Μιχαήλ Γκάλα για τις τροπολογίες στον προπολογισμό που εμπίπτουν σε αρμοδιότητες άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Είναι γενικότερο θέμα. Όπως είπε ο Μιχαήλ Γκάλα, ήταν εξαιρετικά πολλές 21 τροπολογίες από 129 για γραμμές του προπολογισμού που δεν είναι της άμεσης δικής μας αρμοδιότητας. Ε, είναι κυρίως της ΔΕΒΕ και της ΛΥΒΕ. Κατανοώ ότι υπάρχουν επικαλύψεις ε, σε σχέση με τη δική μας δουλειά και άλλα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών και αν μη τι άλλο, όταν ζητάμε να αλλάξουν ποσά, ε, θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση με τις ίδιες επιτροπές. Κατανοώ επίσης ότι στην αρχή μιας θητείας, μιας κοινοβουλευτικής περίοδου, μπορεί να μην γνωρίζουν ακόμα τα ήθη και τα έθιμα εδώ οι νέοι συνάδελφοι. Γι' αυτό σε συνεννόηση με τον εισηγητή αποφασίσαμε αυτή τη φορά να είμαστε πιο επίκης ε, απαράδεκτες εκρίθησαν μόνο οι τροπολογίες που αφορούσαν αποκλειστικά άλλο ε, αντικείμενο, άλλη επιτροπή. Γιατί το λέω, ε, γιατί την άλλη φορά θα είμαστε πιο αυστηροί για να μην έχουμε προστριβές με άλλες επιτροπές. Ελπίζω του χρόνου να μην επαναληφθεί αυτό. Αυτά είχα να σας πω. Θέλω να δώσω το λόγο τώρα στους κοιόδης εισηγητές, η κυρία Νίνα Γκίλ, ο κύριος Λακουτίνσκι, η κυρία Φωτίγκα και η κυρία Ντεμιρέλ άλλο κανει; Ε, η κυρία Σάντο με την τροπολογία τη. Α, ναι, και η κυρία Σάντο. Ε, Προφανώ μάλλον. Πριν την είναι ή μετά. Όχι, πρώτα εγώ γιατί είμαι σκιώδης συγγήτρια. Ε, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μιχαήλ Γκάλερ, λέει η κυρία Γκίλ, για την παρουσίαση αυτή, την εξαντλητική και όλη τη δουλειά που έκανε. Είχαμε καλή συνεργασία θα ήθελα να τονίσω ένα-δύο θέματα. Πρώτον, θα ήθελα να συζητήσουμε την αύξηση ε, στο θέμα των αποστολών ε, παρατήρησης εκλογών. Η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει την αύξηση αυτή. Υπάρχουν όμως κάποιες ανησυχίες για ένα τμήμα της διαδικασίας και θα ήθελα να το αναφέρω θα παρακαλούσαμε τον εισηγητή να το λάβει υπόψη του στις συζητήσεις για να δούμε πώς θα λυθεί. Διότι υπάρχει το εξή ζήτημα. Τέσσερις είναι οι οργανισμοί μόνο που κάνουν παρατήρηση εκλογών. που αναλαμβάνουν να οργανώσουν όλο το ταξίδι και την παρατήρηση εκλογών. Έχω ακούσει όμως ότι είναι ένα καρτέλ αυτές οι τέσσερις οργανώσεις. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε τώρα είναι πολύ πιο ακριβό ε, από ότι αν το οργανώναμε διαφορετικά. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απολύτως με τις αποστολές παρατηρήσεις εκλογών, απλώς θέλω να το θέσω υπόψη σας. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τις απαράδεκτες τροπολογίες, έχω στο γραφείο μου ε, μερικούς ε, συμβασιούχους και εγώ φταίω για αυτές τις τροπολογίες, για την Ασία για παράδειγμα. Ε, τα βάλα σε λάθος κατηγορία, σε λάθος τίτλο. Σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά εδώ έχει γίνει ένα λάθος. Και το τσέκαρα με την Επιτροπή Ανάπτυξης, ΔΕΒΕΙ, που θα ήταν η αρμόδια, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες τροπολογίες εκεί. Δεν θα μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό. Είναι χρηματοδότηση για την Ασία. Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο Μιχαήλ Γκάλερ, η Ασία είναι η μεγαλύτερη και η πιο πολυπληθής ήπειρο στον κόσμο και το 40% του πληθυσμού ζει κάτω από το ε, ε, ε, όριο των 2 δολαρίων ημερησίως. Είναι η δεύτερη φτωχότερη ήπειρο. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε. Δεν θέλω οπωσδήποτε να εγκριθεί η δική μου τροπολογία, αλλά να έχουμε μια αντίστοιχη προσέγγιση, όπως έκανε με όλα τα υπόλοιπα, να πάει στο σχέδιο προϋπολογισμού να επανέλθουν τα ποσά. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κάνει περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό ε, έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό στην Ασία και θα ενταθεί και με τον εμπορικό πόλεμο είπα Κίνας. Δηλαδή σε αυτές τις κοινωνίες οι πιο φτωχοί πραγματικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, να πληρώσουν την τροφή τους. Τεχνικά δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά πραγματικά σε παρακαλώ να το κοιτάξεις. Γιατί του χρόνου θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Δεν μιλώ για χώρε που ανθούν τώρα. Ε, πρόκειται για τους φτωχότερου των φτωχών που δεν μπορούν καν να τραφούν. Μήπως βρούμε καμία λύση. Και όχι αύξηση στο ποσό που προτείνει η δική μου τροπολογία. Τρίτον, για τα πιλωτικά προγράμματα στα οποία αναφέρθηκες. Έχω απογοητευτεί από αυτή την προσέγγιση. Και το έχω συζητήσει πολλές φορές και βλέπω πολλές φορές πώς αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε τροπολογία, πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Ό,τι έχω φέρει εδώ, εγώ οι συνάδελφοί μου, ε, το αποκρύουν. Μου λένε ναι, μα ε, καλύπτεται από αλλού. Μα δεν καλύπτεται από αλλού. Αυτό που προτείνει η κυρία Σάντος, ας πούμε, είναι κατακαιρματισμένο σε διάφορα σύλλο, ε, στεγανά μεταξύ τους και εμείς προτείνουμε αυτό να ενωθεί κάπου θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τι είναι αυτό που μας απαντάτε ότι καλύπτεται από το Α ή το Β project χωρίς να μπορείτε ποτέ να μας αποδείξετε πώς γίνεται. Ε, που μας δίνουν αυτές τις απαντήσεις αλλά μετά δεν το ελέγχουν και δεν, το επαληθεύουν. Αυτό. Ευχαριστώ Νίνα και... Κοιτάξτε. Πολύ ωραία. Έχουμε περίπου 13 λεπτά που απομένουν. Οφείλουμε να κλείσουμε ακριβώς στις 6.30 ε, κυρία Σάντος. Ε, θα τα πω όλα σε ένα ή δύο λεπτά. Εγώ προτιμώ το πρόγραμμα αυτό να προχωρήσει και να περάσουμε στην ψηφοφορία. Διότι εγώ είχα αρκετές ε, συζητήσεις με ανθρώπους που δουλεύουν στην Επιτροπή και έχω κατανοήσει ποιο είναι το πρόβλημα. Ο καθένας έχει τις δικές του τις ε, αρμοδιότητες και μερικές φορές σε κάποιους δεν αρέσει να υπάρχει έτσι μια ομπρέλα, να υπάρχει μια πιο συνεπής εργασία. Εμείς θέλουμε μια ομπρέλα, καλύτερη λογοδεσία καλύτερη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουμε εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όσον αφορά την αντιμετώπιση της ε, ατιμορρησίας, να υπάρχει μια ομπρέλα, να υπάρχουν ελεγκτικά εργαλεία για τις δραστηριότητες μας, να υπάρχει σωστή αξιολόγηση και να υπάρχει και η ικανοποιητική ε, παρουσίαση της ε, δουλειάς μας. μια ολοκληρωμένη προσέγγιση να υπάρχει στο πρόβλημα. Και όπως είπε και η Νίνα, είναι παράδοση πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει συνεχώς όχι. Εγώ προτιμώ να πούνε ναι, προχωρήστε με αυτό το πρόγραμμα, γιατί πραγματικά είμαι πεπισμένη για την αξία αυτού του προγράμματος. Ευχαριστούμε. Κύριε Λακουντίνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε επίσης ε, τον κύριο εισηγητή, τον κύριο Γκάλερ, πάρα πολύ καλή δουλειά και πολύ καλή συνεργασία μαζί του ε, και εκτιμήσαμε ιδιαίτερα το ότι έγιναν αποδεκτές κάποιες από τις ε, τροπολογίες μας, κυρίως όσον αφορά γλωσσικά θέματα, προστίκες δικές μας για τη μετανάστευση. Το εκτιμήσαμε ιδιαίτερα. Υπάρχουν όμως δύο τροπολογίες που θέλω να τις επισημάνω που για μας είναι σημαντικές, επιμένουμε σε αυτές και λυπούμεθα πάρα πολύ που άλλοι συνάδελφοι δεν συμμερίζονται τις απόψεις μας. 53-50 είναι μία. Εκεί ε, θέλουμε να παγώσουμε τις ε, συντάξεις για πρώην μέλη της Επιτροπής, εκτός αν έχουμε γραπτές δεσμεύσεις ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και οι διορισμοί σε αυτήν θα είναι και με βάση τη διάσταση του φύλου. Ξέρουμε ότι αυτή είναι μια πολύ ε, ριζοσπαστική απόφαση, αλλά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Για δε στεργάξεις αριθμούς. Έχουμε 75% ε, των μεσαίων στελεχών που είναι ε, άνδρες ε, και μόνο στο τέλος στις τελευταίες, ε, στους τελευταίους διορισμούς, 11 από 47 διορισμούς που έγινε, μόνο 11 ήταν γυναίκες. Άρα μόνο το 23%. Μιλάμε για μεγάλη ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα και αυτό το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κυρίως ε, διότι ε, και η υποψήφια της Επιτροπής έχει και αυτή κατανοήσει το πρόβλημα. Ελπίζουμε από αυτού να υπάρχει κάποια ειλικρινία. Και άλλη μία τροπολογία, 5347, που αφορά τα, τους γραφείες συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να παγώσουμε τη χρηματοδότηση αυτών μέχρι να έχουμε γραπτές εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και θέλουμε να εκφράσουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στη δουλειά των γραφείων συνδέσμων, αλλά θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν αυτά τα γραφεία. Ε, δεν έχουμε τακτές ενημερώσεις και θέλουμε να υπάρχει πρόοδος ε, όσον αφορά τη διαφάνεια. Σε γενικές γραμμές πιστεύουμε ότι η γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ ε, είναι μια καλή πρόταση για τον προπολογισμό και προφανώς στηρίζουμε εκείνα όλα που είναι υπέρ των ε, ατομικών δικαιωμάτων, υπέρ των χωρών της Δυτικής, ε, των Δυτικών Βαλκανίων, ε, αλλά σε γενικές γραμμές θέλω να σας παρακαλέσω να λάβετε υπόψη σας τις δύο τροπολογίες στις οποίες αναφέρθηκα. Κύριε Αφωτίγκα, από την ομάδα ECR, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι και βραχνιασμένη γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Μιχαήλ Γκάλερ για την εξαιρετική και τρομακτική σε δουλειά που έκανε παρά το καλοκαιρινό διάστημα. Ε, στη συντριπτική τους πλειονότητα υποστηρίζουμε τις προτάσεις του. Θέλω να πω δύο λόγια μόνο και να ρωτήσω και κάτι ε, τον εισηγητή. Πρώτον, ένα τεχνικό ζήτημα Έχουμε την πρόθεση αύριο να υποστηρίξουμε την προφορική του τροπολογία, είναι προφανές αυτό, και προτείνουμε να ακολουθήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την προπαρασκευαστική δράση και τα πιλωτικά προγράμματα για την καταπολέμηση και την εξάλληψη της ατιμορρησίας. Φυσικά όλοι είμαστε κατά της ατιμορρησίας στο διεθνές δίκαιο, όλοι είμαστε και νομοθέτες και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για γραμμές του προπολογισμού θα πρέπει να παραμένουμε λογικοί στη δράση μας και να αποφεύγουμε επικαλύψεις σε θέματα οικονομικά. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι βαθμολόγησε με η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση αυτή. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω ε, κάποιες αμφιβολίες για τη συγκεκριμένη οργάνωση, ε, όχι ως προς τους ε, σκοπούς που είναι ευγενείς και τους υποστηρίζουμε για την παρατήρηση ε, ε, των εκλογών, αλλά έχουμε και μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για σοβαρή κακοδιαχείριση των ε, κονδυλίων και θα πρέπει να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να μην βιαστούμε να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση αυτών των αποστολών δεδομένης της κατάστασης. Έχουμε κάποιες ανησυχίες και αμφιβολίες για την παρατήρηση των εκλογών, συγγνώμη, για την Ούνρα στην Παλαιστίνη. Αντίθετα, όντω για την παρατήρηση των εκλογών συμφωνούμε. Να δούμε όμως τι γίνεται με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, για, αν δικαιολογείται η αύξηση. Ετέθη ένα ζήτημα που είχαμε θέσει εμείς στις οπολογίες μας, ιδιαίτερα Στην περασμένη θητεία η Επιτροπή, που η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας ε, ΣΕΝΤΕ επισκέφθηκε επανειλημμένα τη Γεωργία και είδαμε πόσο σημαντική ήταν η βοήθεια που δίνουμε εκεί και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χαράξη των συνόρων, την ε, προστασία των συνόρων. Ο ρόλος είναι πολύ σημαντικό εκεί και θα πρέπει να στηριχτεί. Ευχαριστώ. Και πριν ξαναδώσω σύντομα το λόγο ε, στον εισηγητή, η κυρία Ντεμιρέλ από την Ενωτική Αριστερά. Κυρία Ντεμιρέλ, κυρία είπε. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, σύντομα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις τροπολογίες της ΓΚΟΕ. Ε, μπορώ να τα πω με τρεις λέξεις συνθηματικά. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα μέτρα ε, μείωσης των εξοπλισμών, εφοπλισμού και ιδιαίτερα ε, γραμμές από το προπολογισμό που είναι υπέρ του εξοπλισμού και της στρατικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιχαράκωσης, θέλουμε να τις ε, καταργήσουμε. Πολύ σύντομα, περί τίνος πρόκειται βλέπουμε συνεχώς να αυξάνονται οι δαπάνες για το Frontex. Και τις τελευταίες ώρες, δύο-τρία ώρες, συζητάμε πάρα πολύ εδώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το είδαμε το καλοκαίρι, είδαμε τι έκανε η Frontex ότι κάθεται εκεί και ε, απαθώς παρατηρεί τα τεκτενόμενα, το πώς αποθείται ο κόσμος. Ε, θα πρέπει εμείς να καταπολεμήσουμε τις αιτίε της φυγής του κόσμου και ε, αντί να κάνουμε τώρα με το Frontex ε, στρατιωτικοποίηση των εξωτερικών μας σύνορων. Επίσης θέλουμε να μην υπάρχουν δαπάνες έρευνας για τη στρατιωτική έρευνα και το αντίστοιχο ταμείο ε, είναι πολιτικά λάθος και όχι μόνο αυτό, είναι και παράνομο γιατί αντιτίθεται στη συνθήκη, στη βασική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 41 παράγραφος 2. Γι' αυτό τα μέτρα αυτά ε, τα θεωρούμε λάθος με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Και αυτό δεν είναι μια υπόθεση της δικής μας ομάδας, μια εικασία. Ζητήσαμε και νομική γνωμοδότηση και μας το επιβεβαίωσε αυτό. Και ένα τελευταίο προσωπικό σχόλιο, κύριε Γκάλερ. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη δουλειά που κάνατε καλοκαιριάτικα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί είστε αντίθετος με τη δική μας τροπολογία ε, για τη μη διάδοση των πυρηνικών και των στρατιωτικών δαπανών. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είδαμε τώρα τι έγινε με την καταγγελία της σύμβασης, μάλλον της συνθήκης για τα, τους πυράβλους μέσου βεληνικούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, INF. Ε, περίμενα ότι θα υποστηρίζατε αυτή την τροπολογία, γιατί για τα κράτη-μέλη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλους είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε. Άλλος κανείς θέλει το λόγο, όχι ο Μίχαελ Γκάλερ για να κλείσει. Ξανά και θυμίζω ότι σε ένα λεπτό θα τελειώσει η συνεδρίαση κανονικά. Ε, τρία λεπτά λέει εδώ το ρολόι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι ε, ε, για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια από τα ζητήματα. Στα πλαίσια των αποστολών για την παρατήρηση εκλογών υπάρχουν τέσσερις διεθνείς οργανισμοί που φαίνεται καμιά φορά ότι λειτουργούν ως καρτέλ. Φυσικά εγώ είμαι κατά των, μονοπολι... των καρτέλ και θα πρέπει και κλεισμένο των θυρών να το συζητήσουμε αυτό το θέμα με κάποιους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή μαζί χωριστά για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις και να διασκεδαστούν αυτές οι εντυπώσεις. Στη συνέχεια. Για τις δραστηριότητες στην Ασία. Ε, προφανώς δεν μπορούμε εμείς να αντισταθμίσουμε όλες τις περικοπές των Ηνωμένων Πολιτειών ε, από το δικό μας προϋπολογισμό. Αν δούμε παγκοσμίω τα αριθμητικά στοιχεία, αυτό θα ήταν υπερβολικό για μας βλέπουμε η τωρινή κυβέρνηση να κόβει όλα τα καλά που έχουν κάνει προηγούμενε αμερικανικέ κυβερνήσει, Δεν μπορούμε εμεί να του αντικαταστήσουμε όσο ευγενεί και να είμαστε ε, στι προθέσει μα. Για την Ινδία υπάρχει ένα ε, κέντρο επιχειρηματικό Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας ε, υποβλήθηκε αυτή μάλλον εγώ το, το σκέφτηκα θα μπορούσαμε να δράσουμε από εκεί σε ό,τι αφορά το θέμα της ατιμορρησίας Θα δούμε πώς θα πάει αύριο στην ψηφοφορία. Επί της ουσίας, θα μπορούσα ενδεχομένως να το υποστηρίξω. Έχω όμως την εκτίμηση ότι ακόμα και εμείς να το υποστηρίξουμε, θα καταψηφιστεί από την Επιτροπή Προπολογισμών. Ε, αλλά αυτό θα το δούμε. Επειδή κυκλοφορούν διάφοροι ανατρεπτικοί πολιτικοί σε υψηλά αξιώματα, ε, δεν χρειάζεται να βάζουμε και εμείς ανατρεπτικές ε, τροπολογίες για την ισότητα και για τις θέσεις σε υψηλά αξιώματα μέχρι να φτάσουμε στην ισότητα των φύλων. Βεβαίως έχετε δίκιο να θέτετε το ζήτημα της ανισορροπίας που υπάρχει ε, ως προς την ισότητα των φύλων. Αλλά νομίζω δεν είναι τώρα ε, χώρος να το κάνετε με τροπολογίες, να το βάλετε στη μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας ε, για να ε, ασκήσετε πίεση, όχι μέσω του προπολογισμού. Φυσικά δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοιε τροπολογίε. Σε ό,τι αφορά τα γραφεία συνδέσμα του Κοινοβουλίου στο εξωτερικό, νομίζω ότι αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά θα δείτε ότι στέλνουν γραπτές εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα πεπραγμένα τους, για τις δραστηριότητές τους. Και όσοι θέλουν να ενημερώνονται μπορούν να ενημερώνονται και να ε, κάνουν και ερωτήσεις ενεργά και για στην καθημερινή δουλειά, αν έχετε μια ε, ε, ιδιαίτερη πληροφορία να μάθετε συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την όνρα και την αύξηση του προπολογισμού, για την ενίσχυση για τους πρόσφυγες. Διάβασα τις κατηγορίες για τη διασπάθηση χρημάτων, για πολύ ακριβά ταξίδια κτλ. Αυτά θα πρέπει να ε, ελεχθούν σε βάθος, αλλά προτιμώ να το γράψουμε πρώτα στον προπολογισμό και από εκεί και πέρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα κοιτάξει τι μπορεί να κάνει και αν υπάρχουν ε, ε, και ζητήματα κακό διαχείρισης και σε περίπτωση που αυτό επαληθευτεί φυσικά θα πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Για τη Frontex τώρα. Αν δεν θέλουμε εμείς ως δημόσιες αρχές από τα κράτη-μέλη να αποσύρουμε την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα και να τα αφήνουμε σε ιδιώτες. Ε, πρέπει να δράσουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το δημόσιο και όχι οι ιδιώτε. Ε, δεν μπορούμε ταυτόχρονα να μειώνουμε τον προπολογισμό του Frontex και όλε οι άλλε δραστηριότητε, οι πιο μακροπρόθεσμε για τη μείωση ε, των αιτίων ε, που διώχνουν τον κόσμο. Προφανώ συμφωνώ, αλλά αυτά είναι πιο μακροπρόθεσμα. Δεν χωράνε στον ετήσιο προπολογισμό τώρα ε, που συζητούμε για το Frontex. Εγώ θα έτεινα να μειώσω τον προπολογισμό, το αντίθετο. Και δεν υποστηρίζω την προσέγγιση σας αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ Μιχέλ Γκάλερ. Ε, αυτά είναι τα σχόλιά σας. δεν έχετε τίποτα άλλο, να κηρύξουμε το πέρας της ε, συνεδρίασης πάνω κάτω στην ώρα μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9, γιατί έχουμε κάτι ψηφοφορίες. Ε, καλό σας βράδυ στις Βρυξέλλες.